Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας προτείνω. Όπως θα είδατε, το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, διάταξη σήμερα είναι η, συνάντηση με την Πολωνική Προεδρία. Θα ήθελα να καλωσορίσω την Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ε, είναι μια συνήθις ε, συνάντηση. Στην αρχή κάθε προεδρίας. Έχουμε τέτοιου είδους συναντήσεις. Θα ήθελα να δώσω στην Υπουργό όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο για να παρουσιάσει τις προτεραιότητες της ε, Πολωνικής Προεδρίας και μετά θα κάνουμε μια συζήτηση. Να καλωσορίσω λοιπόν την Υπουργό Μπιενκόφσκα και θα ήθελα να της δώσω το λόγο. Είναι υπεύθυνη για την περιφερειακή ανάπτυξη ε, και της δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερη ευχαρίστηση να σας παρουσιάσω σήμερα τις προτεραιότητες της Πολωνικής Προεδρίας για την πολιτική συνοχή και την περιφερειακή πολιτική. Η πολιτική συνοχής θα απασχολήσει σημαντικά την Πολωνική Προεδρία αυτό το εξάμεινο. Θέλω να σας πω ότι η Πολωνική Προεδρία έχει μία σειρά προτεραιοτήτων και θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσει να αναπτύσσεται να αναπτύσσεται μέσα από την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την βελτίωση της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες. Τον Ιούνιο παρουσίασε η Κομισιόν για το ε, πολιετές, μια ανακοίνωση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μετά θα εκπονήσει και τα νομοθετικά πακέτα για τα εφαρμοστικά μέτρα του πλαισίου αυτού. Εμείς ε, θεωρούμε ότι η πολιτική συνοχή είναι θεμελιώδης και θα λειτουργήσει ως μοχλό σε όλα αυτά τα μέτρα. Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μπει στην πορεία της ανάπτυξης. Πρέπει να προσεγγίσουμε τους στόχους της Ευρώπης 2020. Η πολιτική συνοχή θα αποτελέσει ένα βασικό στοιχείο της Πολωνικής Προεδρίας Συγγνώμη, αλλά μου έχει έρθει ένας γλωσσοδέτης, λέει ο υπουργό. Μου είπανε να μιλάω αργά. Χρειαζόμαστε μια ισορροπημένη χωροταξική πολιτική στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η πολιτική συνοχή είναι το καταλληλότερο μέσο για την προσέγγιση των στόχων της Ευρώπης 2020. Πρέπει να βρούμε λύσεις ούτως ώστε αυτή η πολιτική να μετρηθεί στο τέλος στα αποτελέσματά της. Πρέπει να έχουμε διαρθρωτικές δράσεις προς τις διάφορες περιφέρειες. Η συζήτηση για την πολιτική συνοχής είναι μια συζήτηση που κρατάει εδώ και τέσσερα χρόνια θα ήθελα να ευχαριστήσω όμως το προηγούμενο την προηγούμενη Τρόικα που βάλανε όλα τα, τα, θέματα επιτάπητος και προετοίμασαν μία ουσιαστικότατη βάση βάση την οποία θα, στην, επί της οποίας θα εργαστούμε η επόμενη Τρόικα, δηλαδή Πολωνία, Δανία και Κύπρος και θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για όλες τις δράσεις που ανέλαβε μέχρι σήμερα. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω για την έκθεση Μάρκους Πίπερ. Είμαι πεπισμένη ότι με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό το μήνυμα το οποίο στείλατε ότι θέλετε μια ισχυρή πολιτική συνοχής θα βοηθήσετε σημαντικά την Πολωνική Προεδρία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Έχουμε προετοιμάσει ένα σχέδιο στα πλαίσια της Τρόικας, ούτως ώστε οι διαπραγματεύσεις για τους κανονισμούς να γίνουν σύντομα και κυρίως συντονισμένα. Συντονισμένα με τις συζητήσεις εκείνες που γίνονται για τον πολιτικό προπολογισμό. Θα ήθελα να μην έχουμε καθυστερήσεις. Αυτό είναι σημαντικό και για μας και για τις επόμενες προεδρίες. Πρέπει να έχουμε το υλικό για να εργαστούμε. Εμείς έχουμε επεξεργαστεί ένα ιδιαίτερα πλούσιο πρόγραμμα για τις ομάδες των εμπειρογνωμόνων. Τώρα πρέπει να ακολουθήσουν βέβαια και οι κανονισμοί που θα παρουσιαστούν ελπίζουμε τον Σεπτέμβριο όπως είχε προβλεφθεί. Ένα στόχος της Προεδρίας μας θα είναι να καταλήξουμε σε μια γρήγορη συμφωνία ώστε να ολοκληρώνουμε τον προγραμματισμό το συντομότερο και να περάσουμε στην εκτέλεση των μέτρων της πολιτικής συνοχής. Θα ασχοληθούμε με ιδιαίτερα σημαντικές θεματικές εντός του πλαισίου της Ευρώπης 2020. Στρατηγικός προγραμματισμός, αποτελεσματικότητα κλπ. Η ευρωπαϊκή η πολωνική συγγνώμη προεδρία θέλει να είναι αποτελεσματική η πολιτική συνοχής. Στο τέλος θα παρουσιάσουμε έναν απολογισμό των εργασιών μας στις 16 Δεκεμβρίου. Θα θέλαμε τον Δεκέμβριο να μπορέσουμε στις, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων να περάσουμε όλα τα σχετικά μέτρα. Τώρα επανέρχομαι και ξαναλέω ότι πρέπει να σεβαστούμε τις προθεσμίες κυρίως για τους κανονισμούς. Να σας πω ποια θα είναι τα εμπόδια ίσως στην όλη πορεία. Πρώτον, στα πλαίσια της επικοινωνίας. Αυτό το νέο μέτρο, το European Connection Facilities, το το μέτρο αυτό πρέπει να αξιολογηθεί ως προς την προστιθέμενη αξία του. Αν η άμεση διαχείριση θα... Πώς θα γίνεται μάλλον η άμεση διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά, τα μεταβατικά μέτρα. Με τη συζήτηση που είχαμε μέχρι σήμερα, βλέπουμε ότι έχουμε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις στις περιφέρειες εκείνες που βρίσκονται σε μια μεταβατική φάση. Η Γνωρίζουμε γιατί. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το μέτρο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο σημαντικό σημείο, το οποίο ίσως να μην είναι τόσο σημαντικό και τόσο πολύπλοκο, αλλά εξίσου σημαντικό, είναι η δυνατότητα του να υπάρχει μία μεγαλύτερη ελευθερία στο κράτος μέλος να κατανέμει τα κονδύλια των διαφόρων ταμείων. Οι αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να αποφασίζουν για το ποια θα είναι η χρήση των κονδυλίων που χορηγούνται. Τώρα, Ευρωπαϊκή χωροταξική συνεργασία είναι η χωροταξική πλευρά της πολιτικής συνοχής. Μετά έχουμε τη στρατηγική για τις πόλεις, έχουμε την στρατηγική για τις μακροπεριφέρειες. Η Πολωνική Προεδρία προσδίδει ιδιαίτερη σημασία σε αυτά τα προγράμματα μέσα στα πλαίσια της χωροταξικής της ε, συγγνώμη, πολιτικής συνοχής Θέλουμε να έχουμε δίκτυα μεταξύ θεσμικών οργάνων, μεταξύ περιφερειών, μεταξύ των το βασικών πρωταγωνιστών σε τοπικό επίπεδο. Θέλουμε δίκτυα στις παραμεθόριες περιοχές. Θα θέλαμε να εναρμονίσουμε τις αρχές της περιφερειακής συνεργασίας. Θέλουμε να προχωρήσουμε όλες τις πρακτικές συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών. Επίσης, θα κοιτάξουμε να δούμε σε δύο φάσεις πώς θα συντονίσουμε την διαπεριφερειακή συνεργασία και αυτό σε επίπεδο Συμβουλίου. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου θα παρουσιαστεί αυτό το σχέδιο. Νομίζω 22 θα παρουσιαστεί από την Κομισιόν. Και τον Σεπτέμβριο λοιπόν εμείς θα πάρουμε αυτή την έκθεση και θα τις ε, συζητήσουμε για την ε, πολιοδομική και χωροταξική ανάπτυξη θα συνεχίσουμε στην υλοποίηση της εδαφικής ατζέντα της Ουγγρικής Προεδρίας. Και θα μιλήσουμε και για την εδαφική συνοχή στα πλαίσια της Ευρώπης 2020. Θα έχουμε ένα background report και ένα issue paper και αυτά θα συζητηθούν στις ομάδες εργασίας των κρατών μελών, δηλαδή στο Συμβούλιο. Κατά δεύτερο, θα συζητήσουμε τις διάφορες ειδικέ λύσεις που προτείνουμε για τις πόλεις, για την Ήπεθρο και για τη σύνδεση μεταξύ πόλης και Ήπεθρου. Θα συζητήσουμε την πρόταση για το μέλλον των πόλεων και θα συζητήσουμε επίσης και το μέλλον του προγράμματος Ουρμπακτ. Κάτι που θέλω να υπογραμμίσω στην Επιτροπή σας. Θα μιλήσουμε για την εδαφική διάσταση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Θα έχουμε μια σημαντική διάσκεψη η οποία θα γίνει στη Βαρσοβία σχετικά με το θέμα. Έχετε στο τραπέζι σας ένα έγγραφο στο οποίο αναφέρονται όλες οι συναντήσεις που θα γίνουν στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής. Τα πιο σημαντικά όμως συμπεράσματα όλων αυτών των συνεδριάσεων, των συναντήσεων θα αποτελέσουν την βάση της άτυπης συνεδρίασης των Υπουργών και τα συμπεράσματά της στις 25 Νοεμβρίου στο Πόσναν. αυτή η άτυπη συνεδρίαση των Υπουργών θα είναι μια διευρυμένη συνεδρίαση. Θα έχουμε τους Υπουργούς, τους αρμόδιους για την χωροταξία, αλλά μαζί συγγνώμη, με τους αρμόδιους Υπουργούς για την Περιφερειακή Ανάπτυξη και την Πολιτική Συνοχής. Θέλουμε να εργαστούμε γύρω από τις μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Αυτοί οι μήνες ε, της ε, Πολωνικής Προεδρίας θα ασχοληθούν σημαντικά με την εφαρμογή της στρατηγικής για την Βαλτική θάλασσα. Ελπίζω, κυρίες και κύριοι, ότι οι διαπραγματεύσεις που θα ολοκληρώσουμε θα βοηθήσουν η στρατηγική μας να γίνεται όλο ένα και πιο αποτελεσματική. Θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις στην ομάδα των φίλων της Προεδρίας στα μέσα Ιουλίου. Θα συζητήσουμε την έκθεση της Κομισιόν για την εκτέλεση αυτών των στρατηγικών. Και μετά το κείμενο των συμπερασμάτων θα το συζητήσουμε στις γενικές υποθέσεις, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων τον Νοέμβριο. 26 Νοεμβρίου. Για να ολοκληρώσω, θα επανέλθω στην αρχή του λόγου μου. Το πιο σημαντικό σημείο της Πολωνικής Προεδρίας θα είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων των κανονισμών για τις πολιτικές συνοχής. Και αυτό είναι σημαντικότατο. Και αν θέλετε αυτή είναι και η πρακτική διάσταση για το τι θέλουμε εμείς να έχουμε ολοκληρώσει στα τέλη Δεκεμβρίου. Το είπα όμως και πριν. Εμείς προετοιμάσαμε ένα μεγάλο, ένα το πρόγραμμα με επίσημες και άτυπες συναντήσεις και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνεδριάζουμε όλο ένα και περισσότερο για τις πολιτικές συνοχής απαιτώντας αποτελέσματα. Είχαμε την πρώτη συνάντηση και όλες την προηγούμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ και σας να συμμετέχετε σε αυτές τις συνεδριάσεις. Διότι θα είστε ιδιαίτερα σημαντική βοήθεια για μας. Η πολιτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφορά τις τοπικές αρχές αφορά τον καθένα σας και είστε λοιπόν καλεσμένοι όλο το επόμενο εξάμεινο να παρίσταστε σε αυτές τις συνεδριάσεις. Ευχαριστώ κυρία Προεδρεύουσα. Αρχίζει η συζήτηση λέει στα αγγλικά η Πρόεδρος. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Καταρχάς, να εκφράσω την ε, ικανοποίησή μου που ανέλαβε η Πολωνία την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτές τις ε, πολύ δύσκολες συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί η Πολωνία ε, εκπροσωπεί την πολιτική συνοχή και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα αποτελέσει έναν από του ακρογωνιαίου λήθους και μία από τι πιο σημαντικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι καλό λοιπόν που ανέλαβε αυτή η χώρα την Προεδρία, γιατί αυτή είναι η χώρα που πάντα έλεγε ότι η πολιτική συνοχή είναι μία από τι πιο σημαντικέ πολιτικέ. Βέβαια αυτό δεν συνέβαινε πάντα. Οπότε τώρα μπορούμε να έχουμε ε, μια αισιοδοξία. Δεν ξέρω αν μπορώ αμέσως να βομβαρδίσω την κυρία Υπουργό με ερωτήσεις. Ίσως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι για την ε, δουλειά που γίνεται από κοινού με την Κύπρο και τη Δανία. Θα μπορούσαμε ίσως να περιμένουμε ότι και οι δύο επόμενες προεδρίες θα προωθήσουν την πολιτική συνοχή. Δεν ξέρω αν αυτό βέβαια είναι πολιτικά σωστή ερώτηση, αλλά θα ήθελα να μας πείτε δύο πράγματα. Και επίσης, πάντα υπήρχε μια ένταση μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, κάτι που είναι φυσιολογικό σε έναν βαθμό. Αλλά ένας, ένας από τους λόγους, πέραν των διαφορετικών που υπάρχει αυτή η ένταση, είναι ότι δεν υπάρχει σαφής ροή πληροφοριών και ενημέρωση. Η δική μου λοιπόν ελπίδα είναι ότι τώρα θα έχουμε επαφή και ελπίζω να γίνει αυτό και σε πιο μόνιμη βάση, έτσι ώστε να ενημερώνει, να ενημερώνει ο ένας τους άλλους για το τι γίνεται, ο ένας τον άλλον για το τι γίνεται ε, στο Συμβούλιο και εμείς να ενημερώνουμε το Συμβούλιο για το τι κάνουμε εδώ. Και επίσης να σας πω ότι θα πάμε στην Ελλάδα, μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας θα πάει στην Ελλάδα, ο συνάδελφος εδώ δίπλα θα είναι ο πρόεδρος αυτής της αντιπροσωπεία και ο επικεφαλής και θα μπορέσουμε έτσι και από τη δική μας τη μεριά να πούμε ότι θα δώσουμε ε, βεβαίως και σε εσά όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ε, επίσκεψη αυτή. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και στρέφομαι σε εσά, ε, κύριε Υπουργέ, με το εξή ερώτημα. Το σημαντικό για μας είναι το πότε θα ξεκινήσει η δουλειά για τους κανονισμούς. Είπατε ότι ελπίζετε να γίνει αυτό το Σεπτέμβρη. Χτες στο Κοινοβούλιο άκουσα να γίνεται μια συζήτηση ίσως για τον Οκτώβριο ή για τον Νοέμβρη. και άκουσα ότι θα υπάρξει και κάποια έτσι, σχέση και με τη γεωργική πολιτική. Ε, ερώτημα λοιπόν, το πιο σημαντικό είναι το πότε θα ξεκινήσει τελικά αυτή η δουλειά. Ίσως εσείς να έχετε κάποιες περισσότερες προφορίες από την ε, Κομισιόν. Δεν θέλω τώρα να προκαλέσω εδώ τα πνεύματα, αλλά ελπίζω να έχουμε μια σαφή απάντηση για το πότε θα αρχίσει η δουλειά, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό. Όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε, τόσο περισσότερε ευκαιρίε θα έχουμε να είμαστε και επιτυχεί και αποτελεσματικοί. Και όλα αυτά να γίνουν και έγκαιρα. Πότε λοιπόν θα ξεκινήσετε να μα στέλνετε α, έγγραφα τα οποία να αποτελέσουν βάση για τη δουλειά μα, για να μπορέσουμε κι εμεί να το συζητήσουμε από κοινού μαζί σας και ένα ερώτημα ε, εκ μέρους του ΕΛΚ. Ας πούμε ότι οι κανονισμοί είναι έτοιμοι, ας πούμε, για το Σεπτέμβρη. Ας υποθέσουμε. Προφανώς, ε, πάντα υπάρχουν πακέτα νομοθετικών εγγράφων και βεβαίως οι προεδρίες θέλουν πάντα κάποια πράγματα να ολοκληρώνονται, να γίνονται θέλουν κάποιοι φάκελοι να περνούν, να κλείνουν. Ερώτημα λοιπόν προς εσάς κύριε Υπουργέ. Ποια είναι τα θέματα που θέλετε εσείς να ολοκληρωθούν. Ποιε είναι οι αποφάσεις, σε ποιους τομείς θέλετε εσείς να ληφθούν αυτές οι τελικές αποφάσεις. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό και για μας. Γιατί έτσι θα επηρεαστεί και η δική μας δουλειά, το δικό μας χρονοδιάγραμμα. Οπότε αν δεχτούμε ότι οι κανονισμοί θα είναι έτοιμοι το Σεπτέμβρη, ποια θα είναι τα θέματα που θα αποφασιστούν και θα κλείσουν μέχρι το τέλος της Προεδρίας. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και βεβαίως θα ήθελα να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία και βεβαίως σύντομα θα δείτε ότι η συνεργασία με τη δική μας Επιτροπή θα είναι αποτελεσματική και ενεργητική. Οι σοσιαλιστές Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω καταρχά την κυρία Υπουργό για την συνάντηση που είχαμε στη Βαρσοβία με τους εκπροσώπους του Υπουργείου περί κάποιους ε, ε, ευρωβουλευτές από, του, από τη δική μου την ομάδα ε, μπορέσαμε, και με κάποιους ευρωβουλευτές από τη δική μου την ομάδα μπορέσαμε να δούμε τις προετοιμασίες της Προεδρίας και πραγματικά σας είμαστε ευγνώμονε για τις πληροφορίες που μας δώσατε άμεσα απευθείας στη Βαρσοβία. Βεβαίω έχουμε και κάποιε αμφιβολίε και θα ήθελα να φίξω το πρώτο σημείο που είπατε για τα ε, ε, πολυεθνικά χρηματοδοτικά πακέτα. Ξέρουμε ποια είναι η θέση της Πολωνίας ε, και εσείς και ο Πρωθυπουργό έχετε παρουσιάσει τη θέση αυτή. Βεβαίως η Προεδρία τώρα ε, κάνει κάποιες συζητήσει για το πώς τα υπόλοιπα κράτη-μέλη ε, βλέπουν αυτή την ε, πρόταση στα πλαίσια πάντα της ε, πολιτικής συνοχή. Εσείς θεωρείτε ότι οι υπόλοιποι υπουργοί είναι διατεθειμένοι να υπερασπίσουν την θέση που παρουσιάστηκε στην Κομισιόν ή θα υπάρξει κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στο Συμβούλιο κάποια προσπάθεια να περιοριστεί αυτή η θέση. Και το ερώτημα είναι, η Κομισιόν και η δική μας Επιτροπή και όλοι εμείς, πώς μπορούμε να ε, υποστηρίξουμε το τμήμα αυτό, το κομμάτι αυτό του, των πολυεθνικών ε, χρηματοδοτικών μέσων Επίση, το είπε, κάτι άλλο που θέλω να θίξω είναι αυτό που είπε και ο κύριο Όλμπριχτ. Ερώτημα προς το Συμβούλιο. Πότε μπορούμε να περιμένουμε το Συμβουλίο και το Κοινοβούλιο ε, αυτό το νομοθετικό πακέτο. Γιατί τα σχέδια που έχετε αναφέρει ε, λυπάμαι, αλλά δεν θα περάσουν εάν το πακέτο δεν είναι έτοιμο το Σεπτέμβριο. Γιατί τότε η Προεδρία δεν θα έχει τίποτα να κάνει, δεν θα έχει τίποτε άλλο να κάνει στα πλαίσια της πολιτικής συνοχής και αυτό ισχύει και για εμάς. Πρέπει λοιπόν να το έχουμε υπόψη μας. Όταν θα έχουμε αυτό το νομοθετικό πακέτο, τότε θα ξέρουμε έτσι περίπου τι γίνεται, ποια είναι τα θέματα που είναι ενδιαφέροντα, ποια είναι τα θέματα που είναι σημαντικά. Και θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εισαγωγή που κάνετε, γιατί αυτό πραγματικά μπαίνει στην καρδιά των, των συζητήσεών μας, γιατί είχαμε κι εμείς ε, κάποια θέματα με τις διάφορες ε, ενδιάμεσες ε, περιοχές, είχαμε ένα πρόβλημα με την Πολωνία για το ποια είναι η θέση της, υπήρχαν κάποιες απόψεις έτσι, αποκλίνουσες και μετά υπάρχει και το θέμα του ποια είναι η άποψη των υπολείπων κρατών μελών για αυτές ακριβώς τις περιοχές. Όλα τα κράτη-μέλη ή κάποια κράτη-μέλη θα είναι έτοιμα να συμπεριλάβουν αυτές τις περιοχές, τις μελλοντικές προοπτικές της πολιτικής συνοχής. Και το ερώτημα επίσης που τίθεται είναι πότε και πώς θα γίνουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. όλες οι προτεραιότητες που παρουσιάσατε η αναθεώρηση δηλαδή της ε, μακροπεριφερειακής πολιτικής και πώς μπορούμε να την ε, χαράξουμε ε, μέσω συγκεκριμένων προτάσεων για τις μελλοντικέ προοπτικές της πολιτικής συνοχής σίγουρα θέλουν να δώσουν μια μεγαλύτερη δύναμη στις ενδιάμεσες περιοχές. Τώρα είναι, μιλούμε για έτσι πιο γενική διαχείριση αυτών των ε, περιοχών. Δεν ε, δρούμε στόχοθετημένα. Ερώτημα λοιπόν. Βλέπετε να υπάρχει ανάγκη για αλλαγή και θα θέλατε να ενισχύσετε τον ρόλο αυτών των περιοχών και περιφερειών. Και επίσης κάτι άλλο που συζητήθηκε στη δική μας την Επιτροπή και εκ μέρου των σοσιαλιστών, θα ήθελα να σας το αναφέρω. Είναι το θέμα της ενίσχυση του ρόλου των περιφερειών. Τα τελευταία χρόνια όλοι ζητούμε νέες ε, δημοσιονομικές προοπτικές ε, και νέα πολιτική συνοχή για να ενισχυθούν οι περιφέρειες, να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες για να μπορούν να λάβουν αποφάσεις για το πώς θέλουν να δαπανούν τα κονδύλια τους στα πλαίσια βεβαίω τη πολιτική συνοχή. Εσεί έχετε έτσι κάποιο πλάνο για το πώ θα γίνει αυτό στο μέλλον. Επίση, ε, πολιτική για τις, ε, ε, για τις πόλεις, για τους αστικούς χώρους. Η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε προς αυτή την ε, πολιτική επίσης ποια θα είναι, αν θέλετε να μας πείτε. Ε, γιατί αυτά τα θέματα σχετίζονται περισσότερο με το μέλλον και με την πολιτική που θα έχουμε από το 2014 έως το 2020. Αλλά τους επόμενους μήνες ποια είναι τα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με αυτή αυτή ακριβώς ε, την πτυχή. Γιατί υπάρχουν ε, προβλήματα στα κράτη-μέλη. Το ανέφερε και ο κύριος Όλμπριχτ, ε, μίλησε για την επίσκεψη στην Ελλάδα. και εμείς όμως στην Πολωνία έχουμε προβλήματα με, την, με τις δαπάνες για την πολιτική συνοχή. Και ειδικά και για, τους, για τις υποδομές, για τους σιδηροδρόμους. ναι, κλείνω, Πρόεδρε. Και επίσης, θα μπορέσουμε να πλουστεύσουμε τελικά αυτά τα συστήματα ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις δαπάνες των ε, κορδιλίων από το Ταμείο Συνοχής. Και πάλι, Πρόεδρε, ευχαριστώ και ε, συγχαρητήρια στην, πρόεδρο, στην ε, Υπουργό για την παρέμβασή της. Δεν έχουμε όσο χρόνο θέλουμε, οπότε ας μην επαναλαμβάνουμε τις ερωτήσεις που έχουν θέσει άλλοι. Και καλύτερα να αποφύγουμε ερωτήσεις που αφορούν συγκεκριμένες χώρες. Ας μιλήσουμε καλύτερα για την Προεδρία γενικώ. Ε, πρόσωπος του Άλτε τώρα. Εγώ θέλω από το λόγο εκ μέρους των φιλελευθέρων σήμερα, αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς, πρέπει να πω, κυρία Πρόεδρε, Ναι, θα μιλήσω για τους συντονιστές, εκ μέρους των συντονιστών, ε, των φιλελευθέρων. Πρέπει να είμαι πάρα πολύ σύντομο παρά το γεγονό ότι αυτά που ακούσαμε ήταν αρκετά. Τέσσερα σημεία θα ήθελα να θέσω. Πρώτον, έχουμε αποστείλει επιστολή ε, στον Επίτροπο και το ίδιο ερώτημα θα θέσω και σε εσά, ε, κυρία Υπουργέ, επειδή εκπροσωπείτε την Πολωνική Προεδρία έχει να κάνει με το ε, πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και την πολιτική συνοχής. Αν δούμε τις συγκρίσιμες τιμές για το 2016... Ο τίτλος 1β που έχει να κάνει με τη συνοχή έχει μια αύξηση του, της τάξης του 5,9%. Σχεδόν 6% δηλαδή άλλη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιφάσκει με την πρόταση αυτή γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι μέχρι τώρα ήταν, υπήρχαν, μιλούσαμε για περικοπές 4% για να μπορέσουν να απορροφηθούν τα κονδύλια σε επίπεδο χωρών Δηλαδή αν είχαμε ένα ΕΠ 100 εκατομμυρίων, 4 εκατομμύρια για παράδειγμα στη χώρα μου, ε, θα ήταν το ποσό που θα έπρεπε να απορροφήσουμε από τα κονδύλια που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα λέτε να το μειώσουμε σε 2,5%. Και αυτό αντιφάσκει με την, με την όλη κατάσταση. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνετε περικοπή στη συνοχή, αλλά μιλάτε για αυτή την αύξηση του 5,9%. Δεύτερον, συνήθως ε, στις ε, προτάσεις ε, δεν υπάρχουν ε, και επεξηγήσεις. Ε, στο νέο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο για τη Γεωργία υπήρξε μια αύξηση τη τάξη του 1 τρίτου. Εδώ για τη μεταβατική περίοδο προτείνεται να παραμείνουμε με τα υπόλοιπα 2 τρίτα. Από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί 2, 3, 4, 5 ή 6% διότι έχουμε μηχανισμούς σταδιακής κατάργησης ε, και δεν καταλαβαίνουμε πολύ καλά όλο αυτό το μαγείρεμα με τα ποσοστά. Γιατί αυτό που χρειαζόμαστε είναι πραγματικά μια εξήγηση αν γίνει η αντικατάσταση των μηχανισμών ε, σταδιακής κατάργησης με τους μηχανισμούς για τη μεταβατική περίοδο συν τα δύο τρίτα των κονδυλίων που αφορούν τις μεταβατικές αυτές περιοχές, θα ήθελα να μου εξηγήσετε τι νόημα έχει το 5% του ε, επίγοντος αποθεματικού. Γιατί εσείς λέτε το 5% να μην καταβληθεί κατά τη διάρκεια της απορρόφησης. Λέτε ότι θα είναι ένα αποθεματικό και ότι στο τέλος όταν η χώρα θα έχει εκπληρώσει πλήρως ε, τις υποχρεώσεις της, το 5% επιπλέον θα καταβληθεί στην τελική πληρωμή. Όμως αυτό δεν ισχύει. Ε, δεν καταλαβαίνω λοιπόν τις ε, συνθήκες υπό τις οποίες το 5% αυτό δεν θα καταβληθεί. Πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εσείς ε, θα, ε, υποβάλλετε, θα υποβάλλετε προτάσεις για τις καταβολές των πληρωμών το, της συνοχής και πώς θα συνδεθεί αυτό με το δυναμικό απορρόφησης. Είναι τόσο διαφορετικό το δυναμικό απορρόφηση ε, στι 27 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση που χρειαζόμαστε ε, επιγόντω να μας εξηγήσετε τι εννοείτε. Μάλιστα, η κυρία Σρόντερ για τους πράσινους. vielen Dank. Ε, vielen Dank. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Υπουργό για το θάρρος που επέδειξε θα έχετε να αντιμετωπίσετε πολλές δυσκολίες να βρείτε συμφωνία στο Συμβούλιο και κατά πάσα πιθανότητα θα έχετε και λίγο χρόνο για να το κάνετε αυτό. Πιστεύετε ότι... Με ακούτε καταρχάς, εντάξει. Ωραία. Έχετε χρόνο, πιστεύετε. Γιατί είπατε δύο φορές ότι είναι σαφές ότι η Κομισιόν το Σεπτέμβριο θα δημοσιεύσει τις ε, προτάσεις. Εμείς υποθέτουμε ότι αυτό θα γίνει αργότερα. Και θα με ενδιέφερε εσείς πώς θεωρείτε ότι θα υπάρξει η θέση του Συμβουλίου τελικά. Γιατί εσείς είστε αυτοί που έχετε τη μοναδική ευκαιρία μέσα σε ένα λογικό έφθετο χρόνο να βρείτε μια συμφωνία. Αν δεν τα καταφέρετε εσείς, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία πριν το 2013. Και γι' αυτό υπάρχει μεγάλη ελπίδα ε, να υπάρξει μέσω της Προεδρίας σας συμφωνία στο Συμβούλιο. Είπατε ότι ήδη έχετε ξεκινήσει να, δουλεύετε πριν την ανακοίνωση των ε, προτάσεων για την επίτευξη α, θέσης του Συμβουλίου. Επίσης, για τις ενδιάμεσες κατηγορίες, για την κατανομή των κονδυλίων, για, την, ε, για το Ταμείο Διασύνδεσης, θα υπάρξει για αυτά τους τομείς ήδη θέση πριν δημοσιεύσει η Κομισιόν α, ε, προτάσεις της. Γιατί αλλιώς δεν θα έχετε πολύ χρόνο αν έρθουν αργότερα οι προτάσεις, ώστε μέχρι τον Δεκέμβριο να έχετε καταλήξει σε μια θέση. Και επίσης, πώς θα καταφέρετε οι χώρες που είναι ε, αυτοί που πληρώνουν ουσιαστικά να βρεθούν σε μια ισορροπία μέχρι τον Δεκέμβριο στην ε, εκπόνηση της κοινής θέσης του Συμβουλίου. Ε, γιατί θα υπάρξουν κάποιες ειδικέ μέθοδοι που θα χρησιμοποιήσετε για να μπορέσετε να φέρετε και τις ε, και τις χώρες αυτές ε, με το, με το μέρος σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Υπουργέ, Χαίρομαι όλους ιδιαίτερο που συναντιόμαστε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να πω ότι η Πολωνία ήταν πάντοτε υπέρο, υπέρμαχος της ε, πολιτικής συνοχής και θυμάμαι την εξαιρετική μας συνεργασία κατά τη διάρκεια της ε, Τσεχικής Προεδρίας και την ε, συνάντηση που είχαμε με εκπρόσωπό σας τότε. Ελπίζω ότι η εμπειρία σας στον τομέα αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να ε, σημειώσουμε πρόοδο κατά τη διάρκεια της Πολωνικής Προεδρίας. Αναφέρατε στην εισαγωγή σας τη σημασία της αστικής διάστασης ε, του μέλλοντο της πολιτικής συνοχής. Ε, εμείς πιστεύουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας και γι' αυτό θα ήθελα να σα ρωτήσω πώς προτίθεστε να εμβαθύνετε ε, στην προσέγγιση των εταιρικών σχέσεων σε, στα διάφορα επίπεδα τοπικών και περιφερειακών αρχών από το εθνικό μέχρι το τοπικό επίπεδο προκειμένου αυτή η προσέγγιση εταιρικής σχέσης ε, να υλοποιηθεί υποστηρίζετε τα ολοκληρωμένα προγράμματα για τις πόλεις του μέλλοντος που είναι ουσιαστικά το εργαλείο της συνεργασίας της και θα ήθελα να σας ρωτήσω Μήπως έχετε σκοπό να προετοιμάσετε ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο για τη συγχρηματοδότηση των ευρωπαϊκών αυτών προγραμμάτων. Γιατί όπως γνωρίζετε το ε, μέσο Jessica δεν έχει χρησιμοποιηθεί πλήρως ούτε ιδιαίτερο συχνά και πιστεύουμε ότι πραγματικά αυτό είναι ο δρόμος για το μέλλον. Ε, η άλλη μου ερώτηση αφορά το μέλλον ε, της μακροπεριφερειακής στρατηγικής. Ε, κατά τη Σουηδική Προεδρία αρχίσαμε την προετοιμασία της ε, στρατηγικής Βαλτικής θάλασσας, μετά υπήρξε η αντίστοιχη στρατηγική για το Δούναβι και τώρα μιλάμε για την στρατηγική για τον Ατλαντικό. Εχθές ασχοληθήκαμε με την έκθεση του κυρίου Αλφονσί που αφορά την περιοχή της Μεσογείου και μιλήσαμε και για την περιοχή των Καρπαθίων. Σε ποιο βαθμό εσείς ε, υποστηρίζετε την μακροπεριφερειακή στρατηγική και ποιος είναι ο βασικός δεδομένου ότι η σημασία της έγκυται ε, στην, ε, στο συντονισμό και όχι στη δημιουργία νέων μέσων. Dziękuję Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά πρώτα να κάνω μια γενική παρατήρηση. Όλες ε, οι ερωτήσεις αναφέρθηκαν στην προθεσμία παρουσίαση των σχεδίων κανονισμού. Εγώ θα σας πω το εξή: Εγώ είμαι πεπισμένη ότι τόσο η Προεδρία του Συμβουλίου όσο και η Κομισιόν θα πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν ούτω ώστε αυτό το σχέδιο να καταλήξει όσο το δυνατόν νωρίτερα την Παρασκευή. Είχαμε μία συνάντηση του Συμβουλίου με το Σώμα των Επιτρόπων και συζητήσαμε και με τον αρμόδιο Επίτροπο για την, για την περιφερειακή πολιτική και την απασχόληση. Και όλοι μου είπαν ότι ελπίζουν μέχρι το Σεπτέμβριο να γίνει αυτό. Αυτό μου είπαν οι επίτροποι. Δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει η Πολωνική Προεδρία. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Όλμπριχτ, εμείς έχουμε ένα σαφές φιλοπορία στην Τρόικα με τη Δανέζικη Προεδρία και την Κυπριακή Προεδρία. Και αυτή η συνεργασία λειτουργεί απίθανα. Και σύμφωνα με το φύλλο πορείας, το τρίτο τρίμηνο θα έχουμε συζητήσει τα πάντα Φτάνει βέβαια η Κομισιόν να μας έχει δώσει τις προτάσεις το Σεπτέμβριο. Βέβαια, εγώ φανταζόμουν ότι θα είχαν έρθει τον Ιούλιο, οπότε τόσο το καλύτερο. Θα είχαμε ξεκινήσει ήδη τη συζήτηση από το Σεπτέμβριο. Αλλά εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτω ώστε να κατατεθούν αυτές οι προτάσεις το συντομότερο. Διότι, το ξαναλέω, η πολιτική συνοχής και τα υπόλοιπα είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Πρέπει όμως να ξέρουμε και τι χρήμα θα έχουμε στη διάθεσή μας, διότι άμα δεν ξέρουμε πόσα χρήματα θα έχουμε, δεν ξέρουμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε. Πρέπει όλα αυτά να τα έχουμε, όλα αυτά τα στοιχεία να τα έχουμε για να προχωρήσουμε στους κανονισμούς πάντως. Αυτή η Τρόικα συνεργάζεται πάρα πολύ καλά. Στην αρχή θα εξετάσουμε τα πιο σημαντικά θέματα ό,τι αφορά τον προγραμματισμό. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έναν καλό προγραμματισμό για να μπορέσουμε να περάσουμε στα λειτουργικά προγράμματα. Τα ζητήματα εκείνα που αφορούν στα στρατηγικά πλαίσια, τα Common Strategy Frameworks, ε, τα θέματα επαφής, ε, τα θέματα των διαφόρων προϋποθέσεων και τα θέματα αιρεσιμότητας. Η συνεργασία με την ΡΕΓΙ και με το Κοινοβούλιο είναι θεμελιώδης για μας. Εμείς βασιζόμαστε στην υποστήριξη του Κοινοβουλίου. Την είχαμε εξάλλου, Συναντήθηκαμε με πολλούς από εσά και κουβεντιάσαμε σχετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη βοήθειά σας και είμαι στη διάθεσή σας για να συζητήσουμε ό,τι θέλετε σε αυτό το εξάμεινο. Τώρα, για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και για τον κανονισμό. Ξαναλέω, χωρίς μία πρόταση κανονισμού από την Κομισιόν η Προεδρία, η Πολωνική Προεδρία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και για να απαντήσω στον κύριο Γκουτμάνης, δεν μπορούμε εμείς προκαταβολικά να παρουσιάσουμε μία πρόταση για τις ε, μεταβατικές ε, ε, περιφέρειες πριν έχουμε μία πρόταση στα χέρια μας χωρίς κανονισμό δεν γίνεται τίποτα είναι σαφές ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις που ήρθαν από αριστερά και από δεξιά αλλά πολλές από αυτές τις προτάσεις είναι αντιφατικές μεταξύ τους. Δεν μπορούμε εμείς να συγκρίνουμε περιφέρειες οι οποίες έχουν το 200%, συγκεντρώνουν το 200% του ΑΕΠ και από την άλλη μεριά να, να τις συγκρίνουμε με περιφέρειες οι οποίες έχουν το 75% οι εν μεταβάση περιφέρειες είναι περιφέρειες οι οποίες έχουν περάσει το 75% εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα παραμείνουν σε αυτή την κλίμακα του 75%. Αλλά διαφέρουν σημαντικά από εκείνε που έχουν ξεπεράσει το 90% και οι οποίες είναι σταθερές εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο 90%. Είπαμε είναι πολύ κοντά ίσως μεταξύ τους ως προς το ΑΕΠ, αλλά διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Κυρίως άμα λάβουμε υπόψη μας ότι σε ορισμένες χώρες έχουμε περιφέρειες οι οποίες μόλις πέρασαν το 75% τώρα και είναι περιφέρειες στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η πρωτεύουσα και είναι η πρωτεύουσα η οποία δίνει την οστική δύναμη σε αυτές τις περιφέρειες για να ξεπεράσουν το 75%. Και αυτό είναι τεράστια διαφορά με έναν των περιφερειών που έχουν ξεπεράσει το 90% εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τώρα στον κύριο Βλάσακ για τη συνεργασία και την εταιρική σχέση. Εμείς θέλουμε να συμμετέχουν οι περιφέρειες σε αυτό το συμβόλαιο. Εμείς θα ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό κύριε Βλάσεκ να βρίσκονται οι περιφέρειες εμπλεγμένες όταν μιλάμε εμείς για ε, πολιτική υπέρ των πόλεων ε, για ε, ε πολιτική, αστική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας όπως η Τζέσικα το να δούμε πώς δουλεύει, πώς λειτουργεί το θέμα της αναζωγόνησης των αστικών συγκοινωνιών σε αυτές τις αστικές περιοχές. Και για μας οι αστικές πολιτικές είναι σημαντικότατες, κυρίως η επαφή που έχουν οι πόλοι με τον περιβάλλοντα υπαίθριο χώρο τι επαφές έχει διαμορφώνει η πόλη με την Ήπεθρο. Είναι πάρα πολύ σημαντική για μας η σχέση μεταξύ της πόλης και των ομόρων περιοχών της. Απλούστευση τώρα. Μιλάμε συνέχεια απλούστευση, απλούστευση, απλούστευση, αλλά εδώ και 15 χρόνια κρατάει η ιστορία της απλούστευσης. στις συζητήσεις για αυτές τις προπτικές για τον κανονισμό των δημοσιονομικών μέσων θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αλλάξουμε μερικά πράγματα. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους, ε, για τους οποίους αναφερόμαστε στην απλούστευση. Αλλά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτόν τον προϋπολογισμό και λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς που ήδη λειτουργούν θα κοιτάξουμε να τους ενισχύσουμε. Τώρα πάμε στις μακροστρατηγικές. Ε, Παρουσία, ε, πολύ θίξατε το θέμα. υποστηρίζουμε όλες τις πρωτοβουλίες εκείνες σχετικά με τις διάφορες στρατηγικές σε περιφερειακό και μακροπεριφερειακό επίπεδο. Έχουμε τη στρατηγική για τη Βαλτική, μίλησα γι' αυτό προηγουμένως, μίλησα για τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ, και τις εθνικές πολιτικές είναι πολύ σημαντικοί και οι δείχτες επίσης. Τώρα υπάρχει το και το όμως και το οικονομικό ξέρετε διότι εντάξει να έχει κανείς στρατηγικές μακροπεριφερειακού χαρακτήρα αλλά μετά χρειάζονται και τα λεφτά. Θα μπορούσαμε να έχουμε ναι και τη στρατηγική των Καρπαθίων αλλά όλα αυτά εξαρτώνται από ε, από τη βούληση των περιφερειών, των τοπικών ε, θεσμικών οργάνων, τοπική αυτοδιοίκηση για να επεξεργαστούμε μακροπεριφερειακές στρατηγικές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να ανασύρουμε τα διδάγματα από τη στρατηγική για την Βαλτική είναι το πρώτο μας εγχειρήμα και να δούμε τι, μας, τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί, τι θα πετύχει, τι δεν θα πετύχει. Για να δω τώρα τι άλλο έχω εδώ. Κύριε Γκούτμεν, μιλούσατε για αυτό το απόθεμα 5%. Όπως και με τις μεταβατικές περιφέρειες και άλλα πολλά θέματα, όλες αυτές οι προτάσεις που έχουμε για το πολιετές ε, σχέδιο, ε, όλα αυτά εξαρτώνται από ποια χώρα έρχεται, ε, προέρχεται. Αν ε, τα δούμε όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο όλα αυτά πρέπει να έχουμε συνείδηση για το τι θα παρουσιάσουμε εμείς ως πρώτο θέμα, την αιρεσιμότητα δηλαδή. Εμείς θα πρέπει να μιλήσουμε για διάφορους τύπους αιρεσιμότητας. Η πολιτική συνοχής είναι ένα διαφορετικό θέμα. Ο όταν μιλάμε για μακροοικονομικά ζητήματα. Και όχι μόνο για την αιρεσιμότητα μόνη της, όχι, μιλάμε για αιρεσιμότητα εξάντε και για αιρεσιμότητα εξ Αλλά το Σεπτέμβριο θα έχουμε τους κανονισμούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λέει η πρόεδρος. Δύο λεπτά ο καθένας, διότι δέκα έχουν εγγραφεί. Και για να μας απαντήσει η υπουργό χρειάζεται χρόνος. Λοιπόν, δύο λεπτά ο καθένας. Η, κυρία Μάνερ, συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Υπουργό για την εξαιρετική της παρουσίαση. Έχει υποθεί πολλές φορές ε, ότι έχουμε μπροστά μας ε, μεγάλες προκλήσεις ε, κατά τους ερχόμενους έξι μήνες. Είμαι όμως βέβαιη ότι η Πολωνία θα τα καταφέρει και θα στεφθεί με επιτυχία η Προεδρία της, γιατί όπως είπατε η πολιτική συνοχή είναι πολύ υψηλή προτεραιότητά σας. Θα ήθελα να επιμείνω στην περιφερειακή και διασυνοριακή συνεργασία. Και εσείς το τονίσατε αυτό το θέμα, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός τομέας και χαίρομαι ιδιαίτερα που το τονίζετε αυτό και μάλιστα τόσο πολύ. Είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε τα προβλήματα που έχουμε ε, στο CBC. Ε, το συζητούμε εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Συζητούμε εδώ και πολύ καιρό πώς είναι δυνατόν ε, το NP και το CBC να τα συνδέσουμε προκειμένου να είναι έναν απόσπαστο τμήμα της περιφερειακής πολιτικής. Αναρωτιέμαι αν αυτό είναι τμήμα της, πολιτικής, ε, του προγράμματός σας και αν θα σημειωθεί πρόοδος επ' αυτού κατά τη διάρκεια της προεδρίας σας. Το πρόβλημα είναι με το, με το NPCBC, το πρόβλημα είναι ε, η Ρωσία, γιατί η Ρωσία είναι η μόνη γειτονική χώρα που συμμετέχει στα προγράμματα αυτά και συνεπώς θα είναι πολύ δικαιολογημένο να ε, να συνδυάσουμε και το θέμα της Ρωσίας με τον τίτλο 3 του προγράμματος αυτού. Αναφερθήκατε και σε αυτό το ζήτημα της μακροοικονομίας και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχετε αυτή τη στάση, όπως επίσης και ε, τη στάση σας για το θέμα της Βαλτικής θάλασσας και του σχετικού πιλωτικού προγράμματος να δούμε αν θα υπάρξουν μελλοντικέ εξελίξεις για το θέμα αυτό και αν υπάρξουν θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η άποψή σας και αν έχετε λεπτομερέστερα σχέδια πώς μπορούν αυτές οι μακροπεριφέρειες να συνδεθούν με τον στόχο 3. Έχετε καμία μεταρρύθμιση υπόψη σας. Ο κύριος Σταυρακάκης, δύο λεπτά παρακαλώ. Thank you. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία, κυρία, κυρία Υπουργέ, θα ήθελα και εγώ να ε, σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία. Ε, στην πολιτική ε, συνοχή, θα αρχίσουν διαπραγματεύσεις κατά την δική σας προεδρία ε, για το θέμα το χρηματοδοτικό. Εμείς γνωρίζουμε ως περιφερειακή πολιτική ότι μετά από την έγκριση του πλαισίου αυτού θα μπορούν οι περιφέρειες να συμμετέχουν πλήρως ε, ε, στα περιφερειακά προγράμματα αλλά και στις ε, εταιρικέ σχέσεις επενδύσεων. Αυτό θα έχει ω αποτέλεσμα να μην υπάρχουν πλέον καθυστερήσεις για, στην αρχή κάθε προγραμματικής περίοδου. Μήπως θα μπορούσατε κυρία Υπουργέ να μας ενημερώσετε αν έχετε σκοπό να αναπτύξετε περαιτέρω πρωτοβουλίες ε, για την ε, ενίσχυση των ε, περιφερειών και αν ναι, ποιες είναι αυτές οι πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος, ο Μίκαελ Τόιρερ για δύο λεπτά επίσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, δύο σημεία θα ήθελα να σας αναφέρω. Καταρχάς, τα ταμεία, το, το Διαρθρωτικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής, που είναι ένα πολύ έξυπνο εργαλείο ώστε να έχουμε μακροοικονομική σταθερότητα. Θα ήθελα να ενθαρρύνω την ε, Πολωνική Προεδρία σε αυτό το σημείο να συνεχίζει να πιέζει και να δουλεύει ακριβώς και λόγω της ευρωκρίσης που υπάρχει και του πιο αδύναμου ε, ευρώ και των πιο αδύναμων χωρών στην ευρωζώνη ε, θα μπορούσε όντως ε, να υπάρξει μεγάλη συμβολή στο τομέα αυτό. Ε, τώρα, η απορρόφηση. Σήμερα ελπίζω ότι θα εκδηθεί μια έκθεση για το θέμα των ε, ε, ποσοστών απορρόφησης και των δυνατοτήτων που έχουν τα κράτη-μέλη. Η Πολωνία εδώ, στο παρελθόν, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και εδώ πραγματικά είναι το υπόδειγμα η Πολωνία σε ό,τι αφορά την απορρόφηση κονδυλίων. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω η Πολωνική Προεδρία να αναλάβει μια πρωτοβουλία ώστε αυτές οι περιφέρειες που έχουν δυσκολίες να απορροφήσουν ε, τα κονδύλια να, τα, να τις βοηθήσει για να δουν πώς μπορούν και αυτές να βελτιώσουν τις δυνατότητες απορρόφησης που έχουν. Γιατί αν τώρα μέσα στη μέση αυτής της περίοδου ε, δεν καταφέρουμε να αυξήσουμε την απορρόφηση των κονδυλίων, δεν θα καταφέρουμε τίποτα. Κάντε παρακαλώ κάτι ως προς αυτό. Αναλάβετε έναν ηγετικό ρόλο. Ευχαριστώ. Very much. Ευχαριστώ πολύ, Μαρή Τερέσαντσε Σμιτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την ε, Πολωνική Προεδρία και την ευνοϊκή της ε, στάση για την πολιτική συνοχή ε, η οποία είναι πηγή ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Σας ευχαριστώ που θέσατε στο, στο επίκεντρο της, του προγράμματός σας αυτό το φιλόδοξο σχέδιο για την εδαφική συνοχή. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η θέση σας. Εσείς θέλετε να φανταστείτε έναν ιδιαίτερο κανονισμό που θα δίνει μεγαλύτερη αξία στο στόχο 3 χάθηκε το μικρόφωνο της ομιλήτριας μιλάει χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια συγγνώμη λέει η ομιλήτρια να τα ξαναπώ λοιπόν εγώ ήθελα να αναφέρω τώρα την πολιτική γυτνία εσείς η Πολωνική Προεδρία επικεντρώνει την προσοχή της ε, προς Ανατολάς. Τι γίνεται όμως με τη Μεσόγειο η Αραβική Άνοιξη ήταν ε, μια ιστορική στιγμή. Να δούμε τι θα γίνει όμως το αραβικό καλοκαίρι. Ε, πρόκειται για μια σταυρική στιγμή. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για το τι θα συμβεί. Ευχαριστώ η Κορνέλια Έλς. Ευχαριστώ. Καταρχά, ό,τι καλύτερο στην πολιτική προεδρία. Αυτό που θα ήθελα εγώ σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ που ζούμε και που κυρίω συζητούμε για την πολιτική συνοχή να είναι να υπάρξει στενή συνεργασία. Να γίνουν δηλαδή πολλές συζητήσεις, ε, να γίνουν ε, κάποιες εκδηλώσει, να συμμετάσχουμε όλοι. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν ε, δυνατό, θα ήταν ευθέω μάλλον, γιατί τον τελευταίο καιρό δεν ήταν, τι τελευταίες προεδρίες δεν κατέστη δυνατό και ήταν δύσκολο για μα. Είναι σημαντική λοιπόν η συνεργασία έτσι ώστε να εμπλουτιστούν οι απόψει. Ε, κάτι άλλο σημαντικό είναι το θέμα των ενδιάμεσων κατηγοριών. Είπατε κάποια πράγματα. Σωστό, σωστά είναι αυτά που λέτε και όντω έχετε δίκιο ότι όντω πρέπει να διαφοροποιήσουμε λίγο τα πράγματα μεταξύ των περιφερειών που είναι ε, πάνω από το 75% και τις περιφέρειες που είναι πάνω από το 90% ή τέλος πάντων βρίσκονται λίγο κοντά στο 90%. Νομίζω ότι ε, η διαφοροποίηση λοιπόν εδώ είναι απαραίτητη και θα σας παρακαλούσα εδώ στην Επιτροπή να ε, ασχοληθούμε και εμείς με το θέμα αυτό ενδελεχώς. Δεύτερο ε, θέμα που ήθελα να σας θέξω είναι ότι μιλήσατε για την διασυνοριακή συνεργασία την οποία θέλετε να ενισχύσετε. Ποια είναι τα σημεία που είναι σημαντικά για σας. Εγώ είμαι έρχομαι από μια τέτοια περιφέρεια στα ανατολικά της Γερμανίας, στα σύνορα με την Πολωνία σε αυτή τη γωνιά ζω και θα ήθελα να μου πείτε πού ακριβώς βρίσκονται αυτά τα, αυτές οι τομές που θέλετε να κάνετε. Και επίσης, μιλήσατε για διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ποιες είναι οι δικές σας ιδέες για τα ταμεία αυτά, πώς θα, πώς θα χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Αυτά, αυτά είναι τα ερωτήματά μου. E, <clears throat> ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Με ρωτήσατε για τη συνεργασία για τις μεταφορές. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ... Ε, συγγνώμη για την ε, ε, συνεργασία των τοπικών αρχών κάθε φορά που συζητούμε αυτό το θέμα, μόνο ωφέλη βλέπουμε από την εκπλήρωση του στόχου αυτού. Και πρέπει μία ακόμη φορά να τονίσω ότι πρέπει να δούμε και τις ε, προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί αυτά που μπορούμε να συμπεράνουμε από διάφορες διαπραγματεύσεις και διάφορες συζητήσεις ε, που ακούμε ότι γίνονται προκύπτει ότι τα χρήματα θα δαπανηθούν ε, όχι σε χώρες αλλά σε προγράμματα. Οπότε πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει δηλαδή να τονίσουμε κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων για τις για το σχέδιο των κανονισμών ε, πρέπει να συζητηθεί και αυτό το θέμα γιατί υπάρχει ένα, μια ιδέα αύξησης ε, των κονδυλίων για το θέμα αυτό και φυσικά βέβαια μια τέτοια πρόταση εμείς θα την καλωσορίζαμε, θα μας ικανοποιούσε πλήρως. Τώρα, για τις ενδιάμεσες περιφέρειες. Και αναφέρομαι στην ερώτηση της κυρίας Μάνερ. Μιλήσατε για τα ε, προγράμματα που αφορούν την πολιτική γειτονία. Εμείς καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολα είναι τα προγράμματα αυτά, πόσο δύσκολη είναι η εφαρμογή τους στο πλαίσιο του στόχου 3. Βλέπουμε πόσα πολλά ε, εμπόδια υπάρχουν και πόσα ζητήματα πρέπει ακόμη να επιληθούν πρέπει ενδεχομένως ε, να εναρμονιστούν περισσότερο τα προγράμματα αυτά ή να τα, τα υλοποιήσουμε όπως και τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας παρά το γεγονός ότι από οικονομικής απόψεως ε, ο τομέας είναι πολύ μικρότερος. Είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι της πίτας της ε, περιφερειακής πολιτικής, αλλά για τη δική μας Περοεδρία είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα θα το επανεπισημαίνουμε συνεχώς και οι πρώτες συζητήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω. Τώρα όσον αφορά το ερώτημα για τις ε, ενδιάμεσες περιφέρειες, ε, η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά τις ενδιάμεσες κατηγορίες ε, και αναφέρει ότι οι ενδιάμεσες κατηγορίες αφορούν όλες τις περιοχές ε, από 75% έως 90%. Έχουμε όμως πολύ διαφορετικές περιφέρειες ε, στο πλαίσιο της κατηγορίας αυτής και δεν είναι δυνατόν να τις βάλουμε όλες στο ίδιο καζάνι. Δεν είναι μια πάρα πολύ ομοιογενής κατηγορία. Υπήρξε λοιπόν μια συζήτηση ε, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων προεδριών μάλιστα για το θέμα αυτό και πρέπει να δούμε πώς θα κατανείμουμε τους διάφορους πόρους και τα διάφορα μέσα που διαθέτουμε ώστε, ώστε όλες οι περιφέρειες να αντεπεξέλθουν στο ε, πραγματικό τους δυναμικό. Και θα ήθελα να περάσω τώρα στο επόμενο ερώτημα που αφορά την κρίση και τη σχέση της ε, με την πολιτική συνοχής. Είμαστε πεπισμένοι και νομίζω ότι αυτό αποτελεί πεποίθηση ολόκληρη της Πολωνικής Προεδρίας ε, ότι η πολιτική συνοχής αν μεταρρυθμιστεί σωστά και έξυπνα δεν χρειάζονται άλλωστε και τεράστιες μεταρρυθμίσεις. Μπορεί να αποτελέσει την, η μόνη ευρωπαϊκή πολιτική που μας, ε, θα, θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Γιατί είναι η πολιτική που μας ε, δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων υποδομών ε, μεγάλης κλίμακας αλλά και μικρότερης κλίμακας. Είναι μια πολιτική η οποία μπορεί να χρηματοδοτήσει ό,τι αναφέρεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020. Μπορούμε λοιπόν ε, να τις, ε, ε, όλες αυτές τις ιδέες να τις υλοποιήσουμε στην πράξη μέσω της πολιτικής συνοχής. Έχουμε τους μηχανισμούς στη διάθεσή μας, αλλά πρέπει να είμαστε λογικοί για να μπορέσουμε να είμαστε και επιτυχείς. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι, αποτελεσματικοί, πρέπει να ευθυγραμμίσουμε τα διάφορα μέσα, δεν μπορεί να είναι δωρεάν για όλους, δεν μπορεί να είναι μια πολιτική η οποία θα ε, εφαρμοστεί χωρίς ε, καθόλου κανόνες, πρέπει να ε, πριτανεύσει η λογική, πρέπει να στοχεύουμε με βάση τα αποτελέσματα που θέλουμε να επιτύχουμε. Και αν ε, δει κανείς τις διάφορες χώρες, αν ε, δει κανείς για παράδειγμα την Πολωνία, τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής είναι σαφέστατα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια για την χώρα μου. Όπως είπα, η πολιτική συνοχής μπορεί να είναι ένα μέσο επενδυτικό και χρειαζόμαστε τέτοιου είδους ε, επενδυτική πολιτική, ειδικότερα όταν είναι δύσκολη καιρή, ειδικότερα όταν υπάρχει κρίση. Ειδικότερα συγκεκριμένη πολιτική πολιτική συνοχή μπορεί να αποτελέσει ένα τέτοιο είδου μέσο. Τώρα για το ερώτημα του κυρίου Σταυρακάκη σε σχέση με τι περιφέρειες. Είναι σημαντική εταίρη για την πολιτική προεδρία οι περιφέρειε, Αυτό είναι προφανέ. Θα τι ε, καλέσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ε, βεβαίω και θα συμπεριληφθούν ε, και όταν θα γίνουν οι διαπραγματεύσει για τι συμβάσει των εταιρικών σχέσεων. Λιγότερο από δύο λεπτά, λέει η Πρόεδρος, έχετε κύριε Μάτουλα, για την επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την Πολωνία για την ε, Προεδρία και θα ήθελα να συγχαρώ και την ε, απερχόμενη ε, Ουγγρική Προεδρία για την, τα, σημαντικά της αποτελέσματα στο πλαίσιο μιας περίοδου κρίσης. Ενδεχομένως ε, για λόγους ταπεινοφροσύνης δεν ε, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής ε, στη χώρα της η υπουργό. Ίσως όμως θα έπρεπε να μας πει περισσότερα για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων που ε, εφήρμοσε η, πολιτική, η, η, συγγνώμη, η πολωνική κυβέρνηση είναι πάρα πολύ σημαντική η επιτυχία αυτή και μπορεί να αποτελέσει υπόδειγμα. Είναι μια βέλτιση πρακτική, ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα. Συγχαρητήρια λοιπόν, ε, έχω δει πώς θα καταφέρνετε στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας και του στόχου 3 και πιστεύω ότι θα συνεχίσει η επιτυχία αυτή κατά τη διάρκεια της, πολιτικής, ε, της, Πολων, της Πολωνικής Προεδρίας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους από την Επιτροπή Ρέτζι που σημείωσαν ότι χάρη στα Ευρωπαϊκά Ταμεία και στα Ταμεία Συνοχής η Πολωνία προχώρησε πάρα πολύ. Πρέπει να πω ότι χάρη στην δουλειά της κυρίας Υπουργού αλλά και του συνολικά του Υπουργείου μπορούμε στην Πολωνία να περηφανευόμαστε ότι έχουμε τόσο υψηλό βαθμό απορρόφησης των κορδιλίων. Ε, το ερώτημά μου είναι για τις ε, νέες ε, προ... προοπτικές του προϋπολογισμού πρόσφατα. Έγινε έτσι μια πολύ θερμή συζήτηση σε διάφορους κύκλους, γιατί υπάρχουν δύο σχολές σε ό,τι αφορά το νέο προπολογισμό και το Ταμείο Συνοχής μία σχολή ε, υποστηρίζεται από πολλά μέλη του Κοινοβουλίου και πολλά και λέει ότι θα πρέπει να δώσουμε πολλά ε, κονδύλια για την καινοτομία, για την ανάπτυξη, για τη μείωση των ε, κομπών του διεξουδίου του άνθρακα. Η άλλη σχολή, που είναι η βασική σχολή που εκπροσωπείται μέσα στο Ταμείο Συνοχής, είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι προτεραιότητες που έχουμε θέσει μέχρι τώρα να υπάρξει δηλαδή εξισορρόπηση μεταξύ αναπτυξιακών διαφορών, μεταξύ ε, αναπτυξιακών διαφορών στις διάφορες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορούμε λοιπόν να συνδυάσουμε τις ε, δύο αυτές σχολές που είναι πολύ σημαντικές και οι δύο ανάλογα από το ποια χώρα κατάγεται κανείς. Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν και έχει τεθεί, θα ήθελα να το ξαναπώ. Ακόμη και να έχουμε τον καλύτερο δυνατό προπολογισμό, δεν πρόκειται να έχουμε κανένα αποτέλεσμα αν δεν έχουμε καλύτερου ε, ρυθμού απορρόφηση στα κράτη-μέλη. Και αυτέ οι διαφορέ είναι πραγματικά σημαντικέ. Η Προεδρία σα, λοιπόν πώς θα μπορέσει να εξισορροπήσει, να εξισώσει αυτές τις διαφορές, να μειώσει την γραφειοκρατία, γιατί μιλούμε για πολλές διοικητικές διαδικασίες και για πολλά ε, διοικητικά προσκόμματα τα οποία οδηγούν στο να μην απορροφώνται στο σωστό βαθμό αυτά τα κονδύλια. Ας πούμε, ε, για το λόγο αυτό η Βρετανική κυβέρνηση μιλάει για μείωση των κονδυλίων στο, mm. ή της συμβολής της στο Ταμείο Συνοχής. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις για διάφορα θέματα. Για, για την ε, πολιτική κοινωνική συνοχή πρόκειται για ένα σημαντικό σχέδιο, αλλά θα παίξει το ρόλο του άμα ανεξάρτητα το δούμε έναντι της στρατηγικής 2020, έστω και αν και οι δύο θα πρέπει να συντρέξουν προς τον ίδιο στόχο Ποια είναι η θέση σας για αυτό το θέμα, για την πολιτική γειτονία και συνεργασίας. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μία καλύτερη συνέργεια μεταξύ των διαφόρων ταμείων και έχω κατά νου, γιατί εργάζομαι για τις χώρες ΑΚΕ, μία καλύτερη διάρθρωση μεταξύ του ΦΕΝΤ και του ΦΕΝΤΕΡ έχετε προβλέψει πρωτοβουλίες για προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά ήθελα να πω, υπόθηκαν και άλλα και άκουσα και απαντήσεις που μου άρεσαν. Ο Αλέν Καντέκ. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, γιατί τις ενδιάμεσες περιφέρειες. Αναφέρατε τα κατόφλια και είπατε ότι αυτές τις ε, διάμεσες περιφέρειες θα έπρεπε να τις κλιμακώσουμε μεταξύ του 75% και του 90%. Οι ενδιάμεσες περιφέρειες ε, ε, εντασσόντουσαν μεταξύ του 75% και του 90%. Είχαν μια, έχουν μια ψαλίδα, δεν μπορούμε εμείς να τις κλιμακώσουμε με νέα κατόφλια με μία εκατοστία μονάδα διαφορά, διότι ε, και ο συνάδελφος το είπε, απλούστευση χρειάζομαι. Θα ήταν επικίνδυνο κάτι τέτοιο, θα ήθελα να μου το εξηγήσετε. Ευχαριστώ. Ο Λάμπερτ Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ την ε, Υπουργό για την εισαγωγή της. Η Πολωνία βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης, αλλά η Πολωνική Προεδρία βρίσκεται στην καρδιά της πολιτικής συνοχής. Το ζούμε στο πετσί μας. Τώρα, η βασική ερώτηση που έχω να κάνω αφορά στην προσέγγιση σας που αφορά στην αναθεώρηση και αξιολόγηση της ευρωπαϊκής πολιτικής γυτνίασης. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά συνέπεια εδώ στην Επιτροπή μας έχουμε την αίσθηση ότι θα έπρεπε να ενισχύσουμε την διασυνοριακή συνεργασία σε επίπεδο περιφερειακής πολιτικής. Εσείς πώς τα βλέπετε τα πράγματα, γιατί εδώ σε μας διαφέρουν κάπως οι απόψεις. Ευχαριστώ πολύ. Είναι δύσκολο κανείς να αναφέρει το πολωνικό παράδειγμα. Πρόκειται για ένα παράδειγμα πολιτικής συνοχής σε πολλά επίπεδα. Αλλά ο κύριος Μάτουλα με ρώτησε σχετικά και να του πω το εξή. Τρία πράγματα έτσι μου έρχονται ε, κατά νου και θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Πρώτον, και κάθε χώρα μπορεί να το κάνει, είναι να διαμορφώσουμε την ε, τη διοικητική ικανότητα, την administrative capacity. Δεύτερον, περιφερειοποίηση στην Πολωνία για, και λόγω προβλημάτων στην αρχή δεν λειτουργήσε καλά, αλλά τελικά τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ θετικά, διότι η χρήση των κονδυλίων σε τοπικό επίπεδο λειτουργήσε πάρα πολύ καλά. Και μετά τρίτον δεν θα πρέπει να έχουμε αμφιβολίες και φοβίες ε, την ώρα της ε, λήψης απόφασης. Αν είμαστε πεπισμένοι ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε έναν στόχο πρέπει να τον παλέψουμε. Και να σας πω το εξής. Στην Πολωνία όταν μιλάμε εμείς ε, για την αποτελεσματικότητα ε, και για την ταχύτητα ότι δεν πρέπει να χάνουμε ούτε ένα σεντ, ούτε ένα ευρώ, πρέπει ε, να, για να γίνει κάτι τέτοιο να παλέψουμε για την αποτελεσματικότητα. Η κυρία Βουκατσέσκα μίλησε, με ρώτησε για το νέο προϋπολογισμό. Για αυτήν την αντίφαση, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη αντίφαση δεν υπάρχει αντίφαση στο να μιλάμε, όταν μιλάμε εμείς ε, για την ε, υλοποίηση των στόχων της συνοχής και της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και απ' την άλλη να υποστηρίζουμε εκείνες τις περιφέρειες οι οποίες ε, χρειάζονται κάπως παραπάνω αυτή την πολιτική συνοχής. Αν εμείς παρουσιάζουμε μία εστίαση που να λέει ότι η κάθε περιφέρεια, ακόμη και εκείνη που είναι πιο καθυστερημένη, έχει τη δική της ε, δυναμική. Ε, ε, ας πούμε, δέστε τι έγινε στην Ανατολική Πολωνία, την πιο φτωχή περιοχή της Πολωνίας. Ε, έχουμε ένα σωρό σχέδια που, πάνε, που τίνουν προς την καινοτομία, προς την εκπαίδευση, προς την έρευνα Δηλαδή σημεία που ανταποκρίνονται απόλυτα με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Δεν υπάρχει καμία αντίφαση. Όταν τώρα όταν μάλλον ε, αναφέρθηκα προηγουμένως ε, και το επαναλαμβάνω η Πολωνική Προεδρία θεωρεί ότι η πολιτική συνοχής είναι μια πολιτική που βρίσκεται στο ύπατο επίπεδο των ανησυχιών μας. Είναι μια πολιτική η οποία εφαρμόζεται επί τόπου, είναι μια απτή πολιτική. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να έχουμε κατά νου πάντα αυτόν τον στρατηγικό στόχο της Ευρώπης 2020 και να είναι καθαρό ότι μέσω της πολιτικής συνοχής μπορούμε να την εφαρμόσουμε για το Αναπτυξιακό Ταμείο και το Διαρθρωτικό Ταμείο. Αυτό όλα αυτά θα τα, εμείς θα τα παλέψουμε σε όλη μας ε, την Προεδρία. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς να πετύχουμε είναι ο συντονισμός μεταξύ των διαφόρων ταμείων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετική αυτή η πρόταση για τα στρατηγικά πλαίσια, τα κοινά στρατηγικά πλαίσια, τα οποία θα ένωναν την πολιτική συνοχή με την ε, κοινή αλλιευτική πολιτική και την ε, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το έχουμε καθαρό ο κύριος Καντέκ, χάνεται το μικρόφωνο της, επανέρχεται. Εγώ δεν είπα ότι θέλω να κάνω διάκριση μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, δηλαδή αυτές που έχουν πάνω από 75% και 90%. Εγώ είπα ότι θα πρέπει να αναλογιστούμε τις εσωτερικές συνθήκες μέσα σε αυτήν την κατηγορία, την εσωτερική κατάσταση ε, της κάθε περιοχής. Δεν μιλάμε εμεί για διαχωρισμό αυτής της κατηγορίας στα δύο, δηλαδή να σπάσουμε την κατηγορία 75-90%. Αλλά να σκεφτούμε τι γίνεται μέσα σε αυτές τις περιφέρειες για τη χρήση των απαραίτητων κονδυλίων. Κύριε Βανίστερο για την ε, ε, cross-board nearby. Ε, το ανέφερα προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δήλωση του Κοινοβουλίου. Για αυτήν τη δήλωση συνεργασίας, αυτό το πλαίσιο. Εμένα μου φαίνεται ότι είναι ένα θέμα αρκετά καυτό κυρίως για τις χώρες και τις περιφέρειες που εκμεταλλεύονται περισσότερο αυτά τα σχέδια. Να σας θυμίσω ότι πέρυσι εμείς παρουσιάσαμε ένα non-paper αυτών των πέντε χώρων για τη χρήση και την εκτέλεση αυτού του μέσου. Τον Ιούνιο έστειλαν μία επιστολή έξι χώρες ε, προς την Κομισιόν για την εφαρμογή αυτών των ε, μέσων και την εκτέλεσή τους. Θα προχωρήσουμε πολύ σε αυτές τις συζητήσεις και στόχος μας είναι να συνενώσουμε όλα αυτά τα σχέδια μέσα στο πλαίσιο του στόχου 3 της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ. Περνάω στα αγγλικά και μπορώ να πω ότι εξονότως όλων ότι πραγματικά εκτιμούμε τη δέσμευση που δείχνει η Πολωνική Προεδρία για να προχωρήσει άμεσα στην προετοιμασία της νέας γενιάς τη πολιτική συνοχή γιατί, για μετά την κρίση, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολη η καιρή, οι προκλήσεις είναι πολλέ η, όπως είπε και η κυρία Υπουργό, η Προεδρία είναι έτοιμη να συμβάλλει, όχι μόνο για να μας βγάλει πιο γρήγορα από την κρίση, αλλά για να μας βάλει στο δρόμο της ανάπτυξης που θα ε, οδηγήσει σε βιώσιμες θέσεις εργασίας και θα μας κάνει πιο ανταγωνιστικούς. επίσης, ε, δεσμευόμαστε και εμείς ότι θα συνεχίσουμε να πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει, να υιοθετήσει, να μας παράσχει και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο σύντομα τον νέο, τους νέους κανονισμούς. Δεν βλέπουμε κανένα λόγο να υπάρξει καθυστέρηση στην υιοθέτηση των κανονισμών που ήδη έχουν προετοιμαστεί ε, λέγοντας ότι η δικαιολογία είναι ότι περιμένουμε άλλους, ε, άλλα νομοθετικά κείμενα. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε το Σεπτέμβρη τον κανονισμό για την ε, πολιτική συνοχή και ότι αυτό θα μπορέσει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πάλι σας ευχαριστώ. Και βεβαίω ε, προσβλέπουμε στην αγαστή συνεργασία μα και σε ανταλλαγή απόψεων και στη διαφάνεια του επόμενου μήνε. Σα ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Uh, ξεκινήσουμε τις προφορίες. Ξεκινούμε τις ψηφοφορίες. Ε, δεν μπορώ να φωνάξω πιο δυνατά. Να ελέγξουμε λίγο, ε, να δούμε αν μπορούμε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is open. Could I ask the assistants to leave the... Μπορούν οι βοηθοί, αν θέλουν να συζητήσουν, να βγουν έξω από την αίθουσα. Λυπάμαι, αλλά πραγματικά μας δυσκολεύεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. The vote is open and uh, I would like... Σας παρακαλώ ψηφίστε για να δούμε αν, λειτουργούν, αν λειτουργεί το σύστημα ηλεκτρονικής πληροφορίας. We still lack some colleagues. Could you please put your cards in? Μπορείτε παρακαλώ να βάλετε τις κάρτες σας όλοι και να ψηφίσετε, γιατί ακόμη κάποιοι δεν έχουν ψηφίσει. So we, we close the vote, I understand. I'm sorry. Εντάξει, λειτουργεί λοιπόν το σύστημα. Πάμε στην πρώτη ψηφοφορία. Μίκαελ Τόιρερ. Έκθεση του Μίκαελ Τόιρερ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 Τε, Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 Συμβαστική 8 υπέρ, συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Την 67 θα την ψηφίσουμε. Μπορούμε να πάμε πίσω στην 67, παρακαλώ συνάδελφοι. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 83 και 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβαστική 13. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 90 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, Α, υπάρχει ε, προφορική τροπολογία. Έχει κανείς αντίρρηση με την ε, ε, προφορική τροπολογία. Ωραία. Όπω τροποποιήθηκε λοιπόν 93 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Τροπολογία 98 υπέρ, κατά, αποχέ. εγκρίνεται. Πάμε στα εκτιμώντα. Συμβαστική 1 Συμβαστική 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4 και 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22-23. Υπέρ. Κατά. Ε, να ελέγξουμε νομίζω, να το δούμε ηλεκτρονικά. Για την 22 και 23 άρχεται η ψηφοφορία. The vote Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 27 προς 18. Πάμε τώρα στην τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην ε, απασχόληση. Τροπολογία 9 προφορική τροπολογία. Είναι κανεί αντίθετο με την προφορική τροπολογία. Όχι. Οπότε ψηφίζουμε την 9 όπω τροποποιήθηκε. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Πάμε στη 10. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Πάμε στην 12. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Πάμε στο τμήμα 1 της τροπολογίας 13, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. μήμα 3 της 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Πάμε στη 14 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεκα... Η 15 καταπίπτει. 16 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας α υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε καλύτερα ηλεκτρονικά για το εκτιμώντας α The is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 35 προς 10. Ε, σκέψη Β. Β. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκτιμώντα Σ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Yes. Τέλος προφορίας. Εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στο Μίκαελ. Ε, ε, Πάμε στην ε, Ραμόνα Νικόλ Μανέσκου για τις δημόσιες προμήθειες. 51 τροπολογίες είχαμε και καταφέραμε να έχουμε 10 συμβαστικές προτάσεις. Υπάρχουν κάποιες ακόμα τροπολογίες που πρέπει να τις ψηφίσουμε. Οπότε ξεκινούμε. Συμβαστική 1. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 10, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στη συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 21. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6, την ψηφίσαμε. Την ψηφίσαμε και ήσασταν αντίθετος, αλλά από ό,τι κατάλαβα ήταν λάθος. Τώρα πάμε Ψηφίσαμε την 21, την εγκρίναμε και τώρα πάμε στην 23. Ποιο είναι υπέρ τη 23. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. αποχέ. εγκρίνεται. 34 υπέρ. Κατά. απόχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43, τροπολογία 43 και 44. Έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, το ξέρω ότι κάποιο θα ζητήσει ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε για το δεύτερο τμήμα λοιπόν τη 43 και 44. Closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 26 προς 20. Ε, τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και πάμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονικά, άρχιτη ψηφοφορία. Closed. Πέρας ψηφοφορία εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην κυρία Μανέσκου. We... Και τώρα περνάμε στην ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο Συντονισμού των Οικονομικών Πολιτικών του Μίκαελ Τόρερ. Συμβιβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται σωστά 5 υπέρ κατά απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 11 υπέρ Υπάρχει προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανείς με την τροπολογία αυτή. Οπότε ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 με προφορική τροπολογία διαφωνεί κανείς. Αν όχι, ψηφίζουμε την 17 όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αν θέλετε να ελέγξουμε την τροπολογία 17 όπως τροποποιήθηκε με την προφορική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με συντριπτική ψηφοφορία. 19 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ. Πέρασα την 5. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική... Α, τροπολογία 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το τελικό κείμενο ηλεκτρονικά άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια κύριε Τόρερ. Περνάμε τώρα στην ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας. Ε, την γνωμοδότηση της κυρίας Μόλκοβα μπορούμε να αρχίσουμε. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ. Υπέρ της 26, κατά. 26 λέει η πρόεδρος. Αφού την 27 δεν την, 25 δεν την εγκρίναμε. Ψηφίζουμε την 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στη συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ. Υπέρ της 32 κατά. Αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 47 υπέρ κατά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 αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τώρα κατά τμήματα ψηφοφορία για την 54 το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται περνάμε στην 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 με, με προφορική τροπολογία διαφωνεί κανείς αν όχι την ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 πάμε τώρα 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικός άρχεται ψηφοφορία Πέρας Εγκρίνεται συγχαρητήρια κυρία Σμόλκοβα. Now... Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στο Χέρμαν Βίλκλερ στη γνωμοδότησή του για το κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να αρχίσουμε την ψηφοφορία με τη συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Καλύτερα να ελέγξουμε την τροπολογία 9 ηλεκτρονικός άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 10 με προφορική τροπολογία διαφωνεί κανείς. Αν όχι, την ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε. Υπέρ. Κατά. Συγγνώμη. Δεν σηκώνεται καλά τα χεράκια και δεν καταλαβαίνω. Οπότε να την ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 45. Σε δύο τμήματα ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα. Α, συγγνώμη, το πρώτο τμήμα λέει η Πρόεδρος. Πρώτο τμήμα της 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57. Προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανείς? Αν όχι ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε την 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 68 υπέρ με προφορική τροπολογία. Διαφωνεί κανείς? Ωραία. Ψηφίζουμε τότε την 68 που τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τότε στην 72. Το δεύτερο τμήμα της 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οπότε περνάμε τώρα στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός. άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφε, ο Μίκαελ Τόρε ζήτησε το λόγο μόλις. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ήθελα απλώ ε, να ευχαριστήσω όλους όσους ε, συνεργάστηκαν μαζί μου για τις ε, δύο εκθέσεις που πρώτη φορά ανέλαβα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ τους κοιόδης εισηγητές, τους γραμματείς και τους συμβούλους για τη συνεργασία τους. Μάλιστα, λέει Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε απευθεία στην ακρόασή μας. Αν θέλετε να αποχωρήσετε, παρακαλώ με ησυχία για να μην μας ενοχλείτε. Περνάμε τώρα στο 16, το 16 σημείο τη ημερήσια διάταξης, είναι εδώ και οι δύο προσκεκλημένοι ομιλητέ μας. Είναι μια πολύ σημαντική μήνυα ακρόαση για τη διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, αλλά και για την ε, αστική συνεργασία είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε προσκαλέσει τον Μισελ Παρακαλώ, διακόπτη Πρόεδρος, έχουμε καλέσει τον Μισελ Λομπλέν που είναι διευθυντή προγράμματο του Interreg IVC. Παρακαλώ όλοι οι πολιτικοί σύμβουλοι και οι βοηθοί να ε, κάνουν ησυχία παρακαλώ μέσα στην αίθουσα. Και έχουμε καλέσει και τον Ζων Λου Ντρουμπινί που είναι προϊστάμενος της γραμματείας Ουρμπακτ. Και χωρίς να καθυστερήσω άλλο θα ήθελα να δώσω το λόγο στου προσκεκλημένου ομιλητέ μα. Δεν ξέρω αν θέλετε να καθίσετε εκεί ή να έρθετε εδώ στο βήμα. Καθίστε εδώ, δίπλα μου. Καλημέρα σας. Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, όσο πλησιάζουμε στις διαπραγματεύσεις των κανονισμών ε, ε, που θα γίνουν μετά από τις καλοκαιρινές διακοπές θα έχουμε όλο και περισσότερες μήνυα ακροάσεις για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα τις ιδιαιτερότητες και να ακούσουμε και τα σχόλια για την τρέχουσα περίοδο από όσους είναι υπεύθυνοι για τα διάφορα μέσα που θα θέλαμε να συνεχίσουμε να έχουμε στη διάθεσή μας στο μέλλον και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικές αυτές οι μήνυα ακροάσεις για όλους όσους θέλουν να λάβουν αποφάσεις ε, ε, στο μέλλον με πλήρη ευθύνη και λογοδοσία. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Λομπλάν που θα λάβει το λόγο πρώτος. Έχετε το λόγο. Merci beaucoup, la Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δουλεύει βεβαίω, βεβαίω. Ευχαριστώ. Η παρουσίασή μου θα σας, δείξει, θα, θα, θα σας δείξω ε, μερικές διαφάνειες κατά την παρουσίασή μου. Βέβαια θα δείτε ότι γίνεται στα αγγλικά η, παρου... η προβολή των διαφανειών, αλλά εγώ θα μιλήσω γαλλικά. Δεν ξέρω, θα είναι κάπως καλύτερα το μπλε πάνω στο μαύρο, να δούμε. Έχω διαρθρώσει την παρουσίασή μου σε ε, σε τρία σκέλη. Πρώτον, χαρακτηριστικά του προγράμματος. Δεύτερον, τα αποτελέσματα τα οποία έχουμε προσεγγίσει σε αυτή τη φάση. Και τρίτον, στις ιδέες που τις μελλοντικές ιδέες για την διαπεριφερειακή συνεργασία. Εμείς βρισκόμαστε μέσα στο πλαίσιο της ε, εδαφικής ευρωπαϊκής συνεργασίας πρόκειται για ένα μικρό στόχο 8,7 εκατομμύρια ευρώ 2,52% του συνόλου της περιφερειακής πολιτικής και η περιφερειακή πολιτική είναι 1,01% ε, του συνολικού προϋπολογισμού Έχουμε βέβαια ανταλλαγή καλών πρακτικών, ανταλλαγή στρατηγικών, ανταλλαγή πολιτικών που λειτουργούν από τη μία χώρα στην άλλη, από μία περιφέρεια στην άλλη. Τα 321 εκατομμύρια ευρώ που χρησιμεύουν στη χρηματοδότηση αυτού του προγράμματος μας επιτρέπουν να υλοποιήσουμε πράγματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα. Βλέπετε ότι στα προγράμματα συνεργασίας, δηλαδή τα προγράμματα Interreg, που, έχουμε, που διαχωρίζονται σε τρία κεφάλαια. Το α είναι το πιο γνωστό διότι αφορά σε όλη τη διασυνοριακή συνεργασία 53 προγράμματα που επιτρέπουν να ε, εξαλείψουμε τις δυσκολίες ε, στις παραμεθόριες περιοχές. Μετά έχουμε τα διεθνικά προγράμματα που είναι 13, όπου έχουμε μεγαλύτερο χώρο δράσης ε, και φύγουμε προβλήματα τα οποία δεν λύνονται μέσω των διασυνοριακών προγραμμάτων. Και μετά έχουμε ε, τα, τα διαπεριφερειακά προγράμματα και έχουμε μετά τα άλλα τρία προγράμματα το, ε, που είναι τα προγράμματα σε δύο. αυτό είναι και το πεδίο εργασίας του Interreg 4C. Έχουν μπει και στο πρόγραμμα και η Νορβηγία και η Σουηδία επιπλέον βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι το ποσοστό παρέμβασης είναι πολύ ψηλό διότι μας επιτρέπει να υποστηρίξουμε τα σχέδια κατά 85% των περιφερειών σύγκλησης ενώ των άλλων περιοχών που είναι και, και των πιο πλουσίων υποστηρίζονται κατά 75%. Αυτό το υψηλό ποσοστό συμμετοχής δικαιολογείται από το γεγονός ότι αυτή η συνεργασία απαιτεί μια προσπάθεια δέσμευσης ε, προς τις άλλες ε, ευρωπαϊκές περιφέρειες. Οι 302 εκατομμύρια δε από το ΦΕΝΤΕΡ πάνε κατευθείαν στο σχέδιο για τη διαχείριση του προγράμματος έχουμε ε, μία ε, επιτροπή παρακολούθησης που αποτελείται από τα 29 ε, κράτη, μετά η προεδρεύει η Ρεζόν Παντεκαλέ και μετά μία γραμματεία στη Λίλη, 30 τόμων, 30 τόμων όπου έχουμε 20 άτομα στη Λίλη και μετά έχουμε τέσσερι στο Ροστόκ, στο Κατοβίτσε και μετά στην Βαλένσια. Οι υπόλοιποι πρόκειται για τέσσερα διαφορετικά σημεία πληροφόρησης που εμψυχώνουν το πρόγραμμα στις διάφορες ε, περιοχές. Ε, Έχουμε την Τράπεζα Επενδύσεων του Σλέστι Χολστάιν, η Generalitat, η αυτονομία της Βαλένσια συμμετέχει στο Νότο και ακόμη μία τράπεζα επίσης ανατολικά. Έχουμε μία Managing Authority που είναι η περιφέρεια του Νορ που συνεργάζεται με την Βαλονία για την γραμματεία, όχι μόνο την γραμματεία του 4C αλλά και το 4B το διεθνικό δηλαδή και το πρόγραμμα 4α των δύο θαλασσών. 830 εκατομμύρια ευρώ και η περιοχή του Νόχ Παντεκαλέ είναι και η βασική περιοχή διαχείρισης του στόχου συνεργασίας και 55, απασχολεί 55 άτομα προσωπικό. Ο στόχος του ΙΝΤΕΡΕΚ 4C είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης. Δηλαδή δεν ε, ξαναεφευρίσκει τον τροχό, απλώς διαπιστώνει ε, που, έχουν γίνει, ε, που έχουμε πετύχει πράγματα ή που έχουμε κάνει λάθη για να μην τα επαναλάβουμε και κυρίως ε, θέλουμε να επαναλάβουμε τις επιτυχίες τις οποίες έχουμε καταγράψει στον τομέα της καινοτομίας και στον τομέα του περιβάλλοντος καταρχήν και, ε, και ακολουθούμε τις, ε, τις προτεραιότητες της Λισαβόνας και του Γκέτεμπορκ που είναι η εποχή της σύλληψης του προγράμματος. Έχουμε 14.000 εταιρούς ε, που έχουν μπει μέσα σε 1300 σχέδια. Δεν ήταν όλοι βέβαια, ε, δεν, δεν εγκρίθηκαν όλα τα σχέδια όταν έγινε η προκήρυξη για την επιλογή, αλλά εγκρίναμε 122 από αυτά τα σχέδια όπου συμμετέχουν πάνω από 1.300 οργανώσεις, 82% των ε, περιφερειών του νετς 2 και κάθε ένα από αυτά τα σχέδια, σε κάθε ένα από αυτά τα σχέδια έχουμε 11 εταίρους που συμμετέχουν. Έχουμε, δεσμεύσει, έχουμε δεσμεύσει τα δύο τρίτα του προϋπολογισμού, μας έχουν περισσέψει 100.000 ευρώ για το οποίο θα αποφασιστεί η χρήση του στα τέλη της χρονιάς φέτος ή στην αρχή της επόμενης χρονιάς. Τώρα δεν φαίνεται καλά σε αυτή τη διαφάνεια, αλλά επικεφαλής της θεματικής που ενδιαφέρει τις περιφέρειες είναι η κολόνα η στήλη αριστερά που αφορά στη μεταφορά και το know-how των τεχνολογιών. Η δεύτερη κολόνα είναι η συνεργασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μετά η πράσινη κολόνα αφορά στην ενέργεια και στις μεταφορές δύο τρίτα ενέργεια, ένα τρίτο μεταφορές και μετά έχετε τη δεύτερη πράσινη κολόνα που έχει αρχίσει και ανεβαίνει και αφορά στις κλιματικές αλλαγές. Για τη συμμετοχή χαίρομαι που είναι σαφής αυτή η διαφάνεια διότι ακόμη και αν χρειάζεται να κάνετε προσπάθειες οφθαλμολογικής εξέτασης για να διαβάσετε θα δείτε ότι μεταξύ των 10 διαπιστώνουμε ότι η Ουγγαρία, η Ρουμανία και η Πολωνία βρίσκονται μεταξύ των top 10 ε, συμμετοχή στα προγράμματα. Έχουν την πρωτοκαθερία. Και βλέπουμε ότι λειτουργεί καλά το σημείο πληροφόρησης στο Κατοβίτσε. Μετά έχουμε τους Ιταλούς ε, οι οποίοι μετά από τον Μάρκο Πόλο ή από τον Χριστόφορο Κολόμβο έχουν μία αλλεργία στη συνεργασία. Αυτό είναι γεγονός, γεγονός. Είναι στο τέλος σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα. Μετά έχουμε τρεις ε, βασικούς λιταργικούς στόχους. Πρώτος είναι ανταλλαγή εμπειρίας, δεύτερον συμμετοχή των καλών πρακτικών και τρίτο, η βελτίωση των περιφερειακών πολιτικών. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να καταλάβετε ότι συνεργαζόμαστε με δημόσιους οργανισμούς, είτε καθαρά δημόσιους, είτε οργανισμούς ε, με πλειοψηφία δημοσίου. Στον τομέα της ανταλλαγής εμπειριών αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι στο 99% των σχεδίων έχουμε μια εταιρική σχέση που έχουμε ε, ανακατεμένες ε, περιφέρειες σύγκλησης και περιφέρειες ανταγωνιστικότητας. Και ε, ελπίζω να έχουμε επιτυχίες ε, της, των περιοχών σύγκλησης και να διδαχτούμε από τις αποτυχίες των περιφερειών ανταγωνισμού για να μην τις επαναλάβουμε. Στη μεταφορά των θεμητών πρακτικών, των καλών πρακτικών, είχαμε πάνω από 1.100 καλές ε, πρακτικές ε, στα 41 πρώτα σχέδια. Πρόκειται για κάτι το πολύ, κάπως τεχνικό, αλλά θα βλέπετε συνολικά έχουμε 122 σχέδια τα οποία είναι λειτουργικά Τα αποτελέσματα όμως τα έχουμε από τα 41 πρώτα σχέδια και μόνο με αυτά τα 41 πρώτα σχέδια έχουμε 1121 καλές πρακτικές που έχουμε διαπιστώσει και 29 οι οποίες ε, σε αυτή τη φάση έχουν μεταφερθεί με επιτυχία. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας καλής πρακτικής και μιας πολιτικής. Μια πρακτική για παράδειγμα ας πούμε η ε, το, επιλογή των ε, σκουπιδιών ε, στην βάση ποια είναι η διαφορά της πρακτικής από την πολιτική είναι ότι για την πολιτική χρειάζονται κονδύλια ούτως ώστε να θεσμοθετηθεί νομοθετικά. Τώρα προχωρώ στον κατά πόσο αυτό το πρόγραμμα αποτελεί μοχλό μέσω, ενός, μέσω μιας ειδική τυπολογίας σχεδίων, σχέδια κεφαλαιοποίησης τα ονομάζουμε. Δηλαδή έχουμε διαχειρις μέσα στην ε, εταιρική σχέση έχουμε ε, ε, το θέμα των εφαρμογών των καλών πρακτικών. Βλέπετε ότι στην κάτω γραμμή περίπου 7 εκατομμύρια ευρώ αφιερώθηκαν σε αυτά τα σχέδια κεφαλαιοποίησης και αυτά τα 7 εκατομμύρια ευρώ για το 4C αποτέλεσαν μοχλό, ε, ε, πολλαπλασιάστηκαν δηλαδή επί 82 διότι επηρέασαν κατά την εφαρμογή τους 573 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτος λειτουργικός στόχος, η βελτίωση των πολιτικών τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Βλέπουμε εδώ 50 εθνικές περιφερειακές τοπικές πολιτικές έχουν βελτιωθεί σε αυτή τη φάση μέσω των πρώτων 40 σχεδίων για να σας δώσω λίγο και το μέγεθος για το τι θα μπορούσε να συμβεί στα τέλη του προγράμματος. Έχουμε, στα τέλους του προγράμματος θα έχουμε 200 επιχειρήσεις και με τέτοιου είδους ε, αποτελέσματα βελτιώνουμε 250 περιφερειακές πολιτικές στην Ευρώπη. Σχετικά με το μέλλον της διαπεριφερειακής συνεργασίας η κάθε επιτυχία έχει και την άλλη της όψη. Είμαστε, έχουμε πολλές επιτυχίες σε επίπεδο παρέμβασης. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι έχουμε μαζική ζήτηση και ε, η απασχόληση ε, είναι κάπως ε, δυσανάλογη με τα κονδύλια που έχουμε θα έλεγα ε, επαρκώς δυσανάλογη ούτως ώστε η επίπτωση του σχεδίου να μετρηθεί όχι μόνο κατά την τωρινή περίοδο προγραμματισμού αλλά και πιο πέρα διότι κάθε χρόνο εγώ αναθέτω αυτή τη δουλειά σε ασκούμενους ε, για να μετρήσουν αυτές τις επιπτώσεις αλλά η επίπτωση έρχεται τρία-τέσσερα χρόνια μετά τον προγραμματισμό και είναι κρίμα Κρίμα κυρίως για την Ευρώπη, διότι μη έχοντας τον ε, αρμόδιο της ανάθεσης ε, ε, δεν μπορεί να γίνει πραγματική μέτρηση των επιπτώσεων επί του πολίτη. Και όταν έχουμε τέτοιου είδους προγράμματα στρατηγικά όπως το Interreg 4C, δεν μπορούμε να, και δεν μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα σε άμεση ε, με άμεση μέτρηση πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να το φανταστούμε στο μέλλον. Αν αποφασίσουν τα κράτη-μέλη του Interreg 4C, τότε εμεί θα κοιτάξουμε να εστιάσουμε καλύτερα το στόχος μας που αποτελείται από ε, στην προτεραιότητα δύο από δημόσιους οργανισμούς ε, και για τη στρατηγική ΕΟΥ 2020, Ευρώπη 2020 θα κοιτάξουμε να προτείνουμε να εργαστούμε και για τη διαχείριση γιατί ανταλλαγή ε, για, ως προς τη διαχείριση των ε, περιφερειακών κονδυλίων είναι πολύ σημαντικές, τόσο σημαντικές όσο και η συζήτηση για το περιβάλλον. Τώρα σε αυτές τις διαφάνειες ε, που μπορείτε να τηλεφορτώσετε από το Interreg 4C ή από την ιστοσελίδα. Ε, θα σας δείξω ένα φιλμάκι. Πρόκειται για την επιχείρηση MKW Making Knowledge Work. Ένα σχέδιο μεταφοράς καινοτομίας προς την αγορά και όπου λειτουργεί καλύτερα, ε, λειτουργεί μάλλον σωστά και μπορείτε να δείτε πώς δουλεύει όλο το σύστημα. Ελπίζω ότι δεν θα περάσει σε μπλε σκούρο όπως προηγουμένως και θα μπορείτε να το δείτε. telescopes, contact lenses, remote controls, CDs, lasers, jet engines,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 να ακούσουμε τον κύριο jean Jean-Luc Ντρουγκινί. Ε, χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και φαντάζομαι ότι θα είσαστε και εσείς πολύ πιστικός στην ε, παρουσίαση του, της σημασίας που έχει η δικτύωση. Και σας ευχαριστώ που ήρθατε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Merci de Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας. Και εγώ στα γαλλικά θα μιλήσω. Μετά από το Interreg 4C, εγώ είμαι ο ε, φτωχός ε, συγγενής, για να το πω έτσι. Το Ούρμπακτ είναι ο γιος ε, του Ιντερεγ. Θα το θυμάστε πολύ καλά ότι είναι, μια, ε, είναι αποτέλεσμα μιας κοινοτικής πρωτοβουλίας ε, για, τα υποβαθμισμένε για τις υποβαθμισμένες συνοικίες, για να δικτυωθούν δηλαδή οι συνοικίες αυτές και να επωφεληθούν από το Ούρμπακτ. Το Ούρμπακτ λοιπόν προέκυψε για να ε, μπορέσει να ε, εφαρμόσει τα προγράμματα Urban. Το Urbact 2, στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ξεκίνησε το 2007, τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή μάλλον τα κράτη-μέλη, ε, ενέκριναν μία νέα έννοια της, του αστικού περιβάλλοντος ολοκληρωμένου ε, και βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος. Υπάρχει λοιπόν ε, μία σύγκληση πολιτικής φιλοσοφίας ε, και χρονικής στιγμής μεταξύ της, τους χάρτας της λειψίας που ανέφερα προηγουμένως και του Ουρμπάκτ. Τέσσερα στόχους έχει και ένα όραμα. Τέσσερις στόχους, ανάπτυξη των ανταλλαγών της ανταλλαγής απόψεων, δηλαδή καλύτερη γνώση, ε, δημιουργία ε, γνώσης, ε, διάδοση επίσης των γνώσεων αυτών ώστε και άλλοι πέραν από τους συμμετέχοντες να μπορούν να υποφεληθούν και τέλος υποστήριξη των φορέων της ε, των όσων ε, χαράζουν τις αστικές πολιτικές. Δεν είναι μόνο λοιπόν ε, ένα πρόγραμμα αστικού τουρισμού, είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγών που σκοπό έχει να προωθήσει την ολοκληρωμένη και βιώσιμη αηφόρο αστική πολιτική. Θα εμβαθύνω στη συνέχεια. Να περάσουμε τώρα στα βασικά ε, σημεία τα οποία πρέπει να γνωρίζετε. Πρώτον είναι ένα πρόγραμμα το οποίο καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο, με το οποίο συνδέονται η Ελβετία και η Νορβηγία. Έχουμε αυτή τη στιγμή 29 θεματικά δίκτυα και ένα, μια ομάδα εργασία. Ε, βρισκόμαστε τέλος πάντων σε ένα επίπεδο πολύ μικρότερο από αυτό που σας παρουσίασε ο κύριος Λόμπλα. Προφανώς 330 εταίροι συμμετέχουν αυτή τη στιγμή περίπου 280 ευρωπαϊκές πόλεις, κάτι το οποίο ε, αποτελεί, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πει κανείς και θα επανέλθω και σε αυτό, είμαστε Εκπροσωπούμε το 57% στις ανταγωνιστικές χώρες και 50% ε, για ε, τις υπόλοιπες. Πρόκειται για ε, κάτι το οποίο καταφέραμε να διατηρήσουμε με ιδιαίτερη ακρίβεια. Το Urbact είναι επίσης ε, μια προσπάθεια συνεργασίας ε, με τους διαχειριστικούς φορείς των διαχειριστικών προγραμμάτων. Προσπαθούμε δηλαδή από την αρχή να ζητήσουμε από τις χώρες ε, να συνδέσουν τα δίκτυά τους με τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων αριθμεί το προσωπικό μας 4.500 άτομα ε, άνθρωποι που καθημερινά ασχολούνται με το πρόγραμμα Urbact. Ο προϋπολογισμός του Urbact ε, που είναι κάτι λιγότερο από 70 εκατομμύρια ευρώ, 80% προκύπτει από το ΦΕΝΤΕΡ. Πρόκειται λοιπόν για έναν προϋπολογισμό αρκετά περιορισμένο τώρα. Πώς λειτουργούμε. Λειτουργούμε μέσω ε, διαγωνισμών. Έχουμε κάνει ήδη δύο διαγωνισμούς και περιμένουμε Εν πάση περιπτώσει ε, προετοιμάζουμε, δεν περιμένουμε απλώς ε, τον τρίτο ε, διαγωνισμό και το Δεκέμβριο θα είναι ο τρίτος και ο τελευταίος μας διαγωνισμός. Ελπίζουμε λοιπόν ότι το URBACT ε, θα αφορά ως τότε 450 ευρωπαϊκές πόλεις ε, και θα ήθελα να πω, μπορεί να το καταλάβατε από την προφορά μου, λέει ο μιλητής, ότι ε, το Ούρμπακ θα το διαχειρίζεται η Γαλλία για λογαριασμό όλων των κρατών μελών. Ας περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Βλέπετε εδώ έναν χάρτη. Είναι ο χάρτης ε, όλων των ε, ευρωπαϊκών πόλεων εταίρων του Ουρμπακτ. Ε, θα ήθελα δύο σχόλια να κάνω που για μένα δείχνουν την επιτυχία του προγράμματος αυτού. Βλέπετε ότι οι πόλεις αυτές είναι πολύ καλά ε, ε, γεωγραφικώς κατανεμημένες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, βλέπετε λοιπόν ότι η ανταγωνιστικότητα και η σύγκληση λειτουργούν, παρά το γεγονός ότι δημιουργούν προβλήματα, λειτουργούν όμως. Το πρώτο ήταν αυτό που ήθελα να πω. Το δεύτερο που θα ήθελα να πω για το χάρτη που βλέπετε είναι ότι οι ευρωπαϊκές πόλεις εταίροι του Ουρμπάκτ είναι 17 πρωτεύουσες ευρωπαϊκές, αλλά ε, υπάρχουν και πόλεις 10-15 ε, χιλιάδων κατοίκων. Ε, οι περισσότερες πόλεις όμως έχουν 100 έως 150 χιλιάδες κατοίκους. Τώρα, ποια είναι τα, ποιες είναι οι θεματικές ενότητες για τις οποίες εργάζεται το Urban. Ε, όπως σας είπα, δημιουργήθηκε το 2007 στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Ε, αφορούσε τις πόλεις που δημιουργούν θέσεις ε, εργασίας, όπως επίσης και τις ε, ελκυστικές πόλεις και τις συνεκτικές πόλεις που έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπως η κοινωνική ένταξη ε, και άλλα προβλήματα του αστικού περιβάλλοντος. Αυτά λοιπόν είναι απολύτως σαφή. Θα ήθελα επίσης να σας πω τι ακριβώς είναι το δίκτυο Urbact, τι είναι, το θεματικό δίκτυο Urbact. Είναι μία ομάδα πόλεων που έχει διαλέξει μια θεματική ενότητα, παρουσίασε τη θεματική ενότητα κατά τη διάρκεια ενός διαγωνισμού. Ε, για παράδειγμα, ένα δίκτυο που αφορά τους νέους που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο και την επανένταξη των νέων αυτών. Είχαμε ένα δίκτυο ε, τέτοιου είδους, ε, το οποίο ξεκίνησε η πόλη του Ρότερνταμ. Μπορεί επίσης να αφορά επιστημονικά πάρκα και ε, την δημιουργία τους σε μεσαίου μεγέθους πόλεις. Υπήρξαν τέτοιου είδους δίκτυα. Μερικές φορές λοιπόν ασχολούμαστε με περιβαλλοντικά ζητήματα, άλλε φορές με κοινωνικά. Έχουμε για παράδειγμα και ένα δίκτυο για τα ηλεκτρονικά οχήματα στις πόλεις και την ανάπτυξή τους. Έχουμε τα εναλλακτικά μέσα μεταφορά ε, το ε, πρόγραμμα ε, που έχει ξεκινήσει στην Αυστρία. Επίσης, ασχολούμαστε με τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ιστορικά κέντρα και πρόκειται για θεματικές ενότητες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση. Πρόκειται λοιπόν για μια θεματική ενότητα Έχουμε μια στρατηγική επικοινωνία συγκεκριμένη, έχουμε, έχουμε έναν περιορισμένο ε, προϋπολογισμό όπως σας είπα, ε, μέχρι 70% για τις ζώνες ανταγωνιστικότητας και μέχρι 80% ε, για τις ε, ε, ζώνες σύγκλησης. Μία μικρή διαφορά σε σχέση με αυτά που σας είπε ο Μισελ Λομπλάν για το μέλλον και το ποσοστό χρηματοδότησης που μόλις σας ανέφερα για το δικό μας πρόγραμμα. Ε, ο αντίκτυπος είναι πάρα πολύ μεγάλος για τις ε, ε, πόλεις λόγω της οικονομικής κρίσης και μάλιστα πολλές πόλεις μας λένε ότι να πληρώνουμε αυτό το επιπλέον, αυτό το το 10-20% ε, που απομένει είναι πολύ δύσκολο. Το είδαμε αυτό με ορισμένες ελληνικές πόλεις ήδη και πιστεύουμε, φοβούμαστε δυστυχώς ότι θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα και με άλλες χώρες και άλλες πόλεις και είναι ένα ζήτημα πρέπει να δούμε πώς θα το επιλύσουμε. Η διάρκεια του προγράμματος είναι τρία χρόνια. Έχουμε περιορισμένο αριθμό εταίρων για λόγους αποτελεσματικότητας, γιατί αν ένα δίκτυο έχει πάρα πολλούς εταίρους δεν λειτουργεί ομαλά, γιατί δεν είναι δυνατόν να το διαχειριστεί κανείς. Και κάναμε μία επιλογή όσον αφορά την αριστεία και την ποιότητα. Δηλαδή τα κριτήρια ε, της αξιολόγησης των υποψηφιωτήτων, των προγραμμάτων ε, ε, αγγίζουν την αριστεία. Προσπαθούμε να πάμε όσο το δυνατόν να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο άριστο για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Έχουμε ένα σύστημα λοιπόν πρωτότυπο, ενδεχομένως και μοναδικό η περίοδος 36 μηνών ε, περιλαμβάνει μια περίοδο 6 μηνών ε, σύλληψης και μία περίοδο ε, ανάπτυξης και εμεί ως Επιτροπή Παρακολούθησης μπορούμε να ε, διακόψουμε ένα πρόγραμμα αν ένα πρόγραμμα φαίνεται ότι πηγαίνει με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία και δεν είναι αποτελεσματικό. Αυτό είναι ένας τρόπος ε, για να βελτιώσουμε την ποιότητα των προγραμμάτων. Επιμείναμε και αναπτύξαμε ε, τη μέθοδο Urbact, όπως την, ε, την αποκαλούμε, γιατί θέλουμε να έχουμε ολοκληρωμένα προγράμματα. Προσπαθήσαμε από μεθοδολογικής απόψεως να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Η, αυτό που χαρακτηρίζει το URBACT, το πρόγραμμα ανταλλαγών, είναι ότι κάθε πόλη εταίρος δεσμεύεται να αναπτύξει ένα τοπικό ε, σχέδιο δράσης, πολύ συγκεκριμένο. Δεύτερον, ε, κάθε πόλη εταίρος Ουρμπακτ δεσμεύεται το τοπικό αυτό σχέδιο δράσης να το βασίσει σε αυτό που αποκαλούμε μια τοπική ομάδα στήριξης, δηλαδή μια ομάδα που συγκεντρώνει όλους τους εταίρους τους οποίους αφορά η θεματική ενότητα. Για παράδειγμα, η πόλη του Ρότερνταμ ε, για το θέμα των ε, νέων που εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο. Βλέπουμε ας πούμε διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, θα έχουμε δηλαδή εταίρους που προέρχονται από τον ε, ακαδημαϊκό τομέα, θα έχουμε επίσης ενώσεις οικογενειών αλλά και επιχειρήσεις. Η ιδέα λοιπόν αυτή τη ομάδα στήριξη τη τοπική είναι όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορεί να συμμετέχουν και να δουλεύουν από κοινού για το τοπικό σχέδιο δράση που ανέφερα προηγουμένω. Επίση προσπαθούμε να ε, συνεργαστούμε με τα, τις διαχειριστικές αρχές των επιχειρησιακών προγραμμάτων από την αρχή για να μπορέσουμε να έχουμε και μια χρηματοδότηση γιατί έχουμε μια διαρθρωτική ε, αδυναμία το γεγονός ότι το Urbact δεν έχει, αυτόματο, δεν έχει αυτόματη σχέση ε, με ε, τα επιχειρησιακά προγράμματα, άρα πρέπει να πείσουμε τις τοπικές διαχειριστικές αρχές. Υπάρχει λοιπόν μια έντονη παρουσία της γραμματείας, ε, όπως ε, καταλαβαίνετε, η οποία παρακολουθεί την εφαρμογή των προγραμμάτων με την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει. Έχουμε λοιπόν μια ολόκληρη διαδικασία δημιουργίας γνώσης ε, και σε επίπεδο ε, δικτύων και προγράμματος ε, έχουμε δημιουργήσει τα εργαλεία που μας επιτρέπουν όσο το δυνατόν περισσότερο να περάσουμε από την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε μια δημιουργία γνώσεις ε, που θα μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ε, και πόλεις οι οποίες ε, δεν συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Ουρμπακτ γιατί η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών πόλεων δεν θα είναι ποτέ μέλη του Ουρμπακτ. Επιμένουμε λοιπόν πολύ σε επίπεδο προγραμμάτων αλλά και σε επίπεδο τοπικών σχεδίων. Τι μπορούμε τώρα να παράγουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι Καταρχάς, να ενισχύσουμε όλα τα τοπικά σχέδια δράσης. Ε, ένα πρώτο κύμα 20 τοπικών δικτύων ε, πρόκειται να δημιουργηθούν, δηλαδή 200 τοπικά ε, σχέδια δράσης πρόκειται να ολοκληρωθούν και θα προσπαθήσουν οι πόλεις να τα εφαρμόσουν στην πράξη. Βέβαια πρέπει να κάνουμε και μία σύνδεση αυτή η δουλειά, η διαδικασία που σας παρουσίασα προηγουμένως δεν είναι χιλιάδες σελίδες που κανείς δεν θα μπορεί να διαβάσει αλλά κάποιες, ε, κάποια σύνθεση με συγκεκριμένα στοιχεία ε, σε αυτό το σε αυτή τη διαδικασία που σας ανέφερα προσπαθούμε δηλαδή να έχουμε ε, να τα παρουσιάζουμε ε, σε κάποιες δημοσιεύσεις που ενδεχομένως να είδατε και στην είσοδο της αίθουσας. Ε, προσπαθούμε να έχουμε διάφορα σεμινάρια, έχουμε κάποιες μελέτες, μια μελέτη για παράδειγμα για την ανταπόκριση των πόλεων στην χρηματοοικονομική κρίση. Νομίζω ότι και αυτή είναι διαθέσιμη, αυτή η μελέτη. Ό,τι οργανώνουμε ε, πριν να αποτελεί τμήμα της ε, στρατηγικής της επικοινωνίας μας, θέλουμε να είναι τμήμα της ε, μεθόδου εργασίας μας. Έχουμε μάλιστα και πανεπιστήμια καλοκαιρινά στην Κρακοβία για τα μέλη της, των τοπικών ομάδων στήριξης. Η κυρία Ήμπνερ μάλιστα θα εγγενιάσει το συγκεκριμένο ε, εργαστήριο. Δεν θέλουμε μόνο να γιορτάσουμε την Ευρώπη και να πιούμε ένα ποτηράκι. Θέλουμε να ε, κάνουμε και τη δουλειά μας. Οι συμμετέχοντες όταν λαμβάνουν ε, την πρόσκληση καταλαβαίνουν ότι θα έρθουν στην Κρακοβία, για να δουλέψουν. Και από ό,τι, κατάλαβα, από ό,τι καταλαβαίνετε είναι αυτό ένα σημαντικό τμήμα της σύμβασης που έχουμε μαζί τους. Ποιος είναι ο σκοπός μας. Ε, το κοινό στόχος μας ε, είναι οι χιλιάδες άνθρωποι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Πώς μπορούμε να τους προσεγγίσουμε. Είναι μια τεράστια δυσκολία, όμως αυτό είναι το καθήκον μας. Προσπαθούμε να έχουμε μια ε, ενεργό πολιτική και δεδομένου δεδομένη της, ε, του μεγέθους του κοινού μας ε, βασίζεται στο διαδίκτυο. Έχουμε τον ιστότοπό μας, τον οποίο όλες οι πληροφορίες όλων των δικτύων ενημερώνονται τακτικά. Και περάσαμε, ε, επίσης έχουμε και πολλές συμφωνίες με ιστότοπους σε διάφορες χώρες, στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, 20 τέτοιους ιστότοπους έχουμε, στην Ορβηγία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και πρόκειται για ιστότοπους που αναπαράγουν ουσιαστικά στην ε, ε, γλώσσα ε, της κάθε χώρας τη δουλειά μας. Προσπαθούμε έτσι να προσεγγίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο αυτούς τους ανθρώπους των πόλεων, για να το πω έτσι. Ένα τελευταίο σημείο για την επικοινωνία μας, για το επικοινωνιακό κομμάτι, είναι ότι ένα πρόγραμμα σαν το δικό μας δεν μπορεί παρά να βασίζεται, ειδικότερα για τις γνώσεις, στα κράτη-μέλη. Η γνώση που αναπτύσσουμε πρέπει να ε, χρησιμοποιείται από τα κράτη-μέλη και να διαδίδεται από αυτά. Δεν μπορούμε να φανταστούμε από τις, ότι από, την, ε, από τις Βρυξέλλες ή από τα κεντρικά μας γραφεία ε, θα πρέπει να διαδώσουμε εμείς σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους τα, τις γνώσεις μας. μπορούμε εκπεπιθήσεως νομίζω να πούμε ότι θα διαδίδονται όλα αυτά τα αποτελέσματα και όλες αυτές οι γνώσεις από τα κράτη-μέλη. Και το τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θέσω, μόλις ολοκληρώσαμε ε, την αξιολόγηση, την μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση, ε, την μεσοπρόθεσμη αξιολόγησή μας ε, και θα κάνουμε και βελτιώσεις για τον τρίτο διαγωνισμό που σας ανέφερα. Βεβαίως θα προσαρμόσουμε το πρόγραμμα στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 και θα ήθελα να επιμείνω σε δύο σημεία. Πρώτον, ότι η εμπειρία που έχουμε μας δείχνει πόσο πρακτικό είναι το να έχουμε τοπικές ομάδες στήριξης ε, και να έχουμε, μία επιρροή, να έχουμε μία επιρροή σε σχέση με το πώς εφαρμόζονται τα ε, σχέδια. Και γι' αυτό ζητήσαμε να αυξηθούν ε, οι πόροι για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, για τις ομάδες στήριξης, δεν έχει νόημα να ζητήσουμε από κανέναν ε, ε, να, ε, να, να δημιουργήσει ένα σχέδιο δράσης τοπικό χωρίς να του δίνουμε τους, τα μέσα να το κάνει γιατί χρειάζεται και τεχνογνωσία και πολλά άλλα πράγματα και χρειάζεται και πόρους. Κάτι ακόμη σημαντικό, το οποίο είναι σημαντικό για το εργαστήριο που προσπαθούμε να αποτελέσουμε, Προσπαθούμε να προβληματιστούμε για τη συμμετοχή των ε, ε, εκλεγμένων, των τοπικά εκλεγμένων εκπροσώπων ε, στο δίκτυο. Είναι ένα από τα σημεία που ακόμη προσπαθούμε να επεξεργαστούμε και δεν έχω περισσότερα να σας πω. Ένα ακόμη σημείο αποφασίσαμε στην τελευταία φάση και τον τελευταίο διαγωνισμό να δώσουμε βάση στη βελτίωση της ποιότητας ε, των τοπικών σχεδίων δράσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα συζητήσουμε μεθοδολογικές, ε, μεθοδολογικά ζητήματα, όμως η εμπειρία μας μας δείχνει ότι έχει ένα πραγματικό αντίκτυπο στον κόσμο. Και για να απαντήσω στο ερώτημα της κυρίας Ούμπνερ προηγουμένως, προσπαθήστε να μας πείσετε. Κάθε φορά που εγώ στέλνω τους ε, συναδέλφους μου, ε, εκπροσωπώντας το δίκτυο, μας δείχνουν ότι δουλεύουν, συνεργάζονται, ότι δεν ανταλλάσσουν απλώς απόψεις και προσπαθούν να αναπτύξουν τοπικά σχέδια δράσης και αυτό εμπλουτίζει πάρα πολύ και τις γνώσεις του ενός και τις γνώσεις του άλλου και υπάρχει επίσης και έμπνευση του ενός από τον άλλον. Οπότε έχω συχνά την ευκαιρία να το πω αυτό, οι εταιρείε κάνουν benchmarking σε καθημερινή βάση και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα ήταν ανόητο για τις τοπικές αρχές να κάνουν το ίδιο. Έχουν μόνο κέρδος, θα έχουν μόνο κέρδος από αυτή τη διαδικασία. Οι πόλεις εταίροι του Urbact ε, θα έχουν έτσι μάθει κάτι, θα έχουν πραγματικά ε, μάθει κάτι από, την, ε, από τις ανταλλαγές αυτές και αυτός είναι ο στόχος μας. Ευχαριστώ. Okay. Thank you, Mr. Uh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για, τις για την πολύ χρήσιμη παρουσίαση. Τώρα μπορούμε να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις. Ο κύριος Βανίστελ Ροϊτ έφυγε. Ο κύριος Όλμπριχτ έχει το λόγο. Ζητώ συγγνώμη ε, ο συνάδελφος ε, μου έδωσε τις δύο ερωτήσεις του να τις θέσω εγώ και έχω και μία δική μου ερώτηση. Τα, οι, δύο ερωτήσεις του Λάμπερτ είναι πώς μπορούμε να μεταφράσουμε στο Interreg 4 την, ε, το πώς θα τα ποσοστά και πώς αυτά είναι τόσο υψηλά και πώς μπορούν να, να, να ερμηνευτούν τελικά σε συγκεκριμένα νούμερα, σε συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία. Και επίση το δεύτερο ερώτημα είναι, είναι δυνατόν όλα τα προγράμματα να γίνουν λίγο πιο διαφανή, γιατί υπάρχουν πολλά προγράμματα που βρίσκονται στα πλαίσια του Interreg 4 και έχουν συγκεκριμένα ονόματα, αλλά κάποια αναφέρονται γενικώ ως Interreg. Δεν θα πρέπει να είναι λίγο πιο σαφή τα πράγματα. Κάθε πρόγραμμα είναι ευρωπαϊκό Interreg ούτως ή άλλως. Και δίπλα να αναφέρεται και ποιο είναι το περιεχόμενο του κάθε προγράμματος. Και το δικό μου το ερώτημα. Και στι δύο, ερώτη, και δύο παρουσιάσεις, συγγνώμη, είδα πως ε, με τα συμπεράσματα των δύο ομιλητών ε, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις ε, σχέσεις μας με τις διαχειριστικές αρχές αυτών των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Εάν και στις δύο προτάσεις προτείνεται αυτό, ε, σημαίνει ότι κάπου κάτι λείπει για να ε, παρουσιάζεται ως πρόταση. Είναι κάποια δυναμία αυτό ή απλώς είναι μια πρόταση για το μέλλον. Δεν είναι το ίδιο, γιατί αν θέλετε, αν θα θεωρήσουμε δυναμία, πάνε να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Είναι άλλο αυτό και άλλο να το παρουσιάζουμε ως κάτι πιθανό για το μέλλον. Οπότε πώς ακριβώς πρέπει να το μεταφράσουμε εμείς αυτό. Εφόσον το χρειαζόμαστε, πάει να πει ότι δεν υπάρχει. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Κέλλη. Ε, thank you very much for... Ε, Ευχαριστώ. Πολύ σαφής η παρουσιάση σας. Κάποια σχόλια και κάποια ερωτήματα. Πρώτον, είπατε ότι από εδώ και μπρος θα πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια της στρατηγικής 2020, γιατί πάνω σε αυτό θα κρυθούμε. Αλλά θα επιλέξουμε τους στόχους μας ή όχι για την στρατηγική 2020. Τώρα, είπατε ότι κάποιες περιοχές αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χρηματοδότηση. και μπορεί μόνο να διαθέτουν το 10 ή το 20% ή ακόμα μικρότερο ποσοστό από αυτό. Οπότε εγώ σωστά συνάγω ότι μπορούμε κάποιο, μια ε, χρηματοδότηση να τη χρησιμοποιήσουμε αλλιώ για μία περιοχή και αλλιώ για μια άλλη. Και αν δεν επίπτουν στα πλαίσια τη χρηματοδότηση, το πρόγραμμα αυτή πώ θα το εφαρμόσουν. Δεύτερον, η επόμενη πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι τέλος του έτους. Υπάρχει πιθανότητα να συμβάλλουν και άλλες ε, περιοχές στα προγράμματα αυτά και αν ναι, πώς ακριβώς το διαχειριστείτε. Ευχαριστώ. Okay. Mr. Hall. Ε, sorry, just Α, και άλλο ένα σχόλιο. Συγγνώμη, συγγνώμη. Άλλο ένα σημείο. Είπατε ότι τελειώνει το πρόγραμμα μετά από 36 μήνες. Μιλούμε για τη στρατηγική 2020 υπάρχει νόημα να, να τελειώνει αυτό μετά τους 36 μήνες, ενώ θα έπρεπε ουσιαστικά να τρέχει μέχρι το 2020. Ε, Ευχαριστώ. Ερώτηση για τον κύριο Λάμπερ. Ρωτώ. Ποια είναι τα κριτήρια για τη χρηματοδότηση των σχεδίων Interreg Υπάρχει μία επιτροπή επιλογής για τα σχέδια. Και πώς θα κρίνουμε τα σχέδια. Αυτό ισχύει για όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, όποιες και να είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. π.χ. διαρθρωτικές δυσκολίες, νησιά, μικρά νησιά, κλπ. Μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στη χρηματοδότηση των, των σχεδίων Ιντερνετ. Άλλος κανένας. Παρακαλώ. Okay. Um... Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους κυρίους Λαμπλάν και Ντομπινί που ήρθαν να με συναντήσουν σήμερα. ερώτηση που αφορά και στους δύο. Η ζήτηση των σχεδίων, οι αιτήσει είναι πολύ περισσότερες από ό,τι δυνατότητες επιλογής και ε, αυτό δημιουργεί πολύ περισσότερο, μεγάλο φόρτο εργασίας αλλά και η απόρριψη δημιουργεί απαγοήτευση κλπ. Πώς θα αντιμετωπίζετε αυτό. Συζητήσαμε κατά πόσο θα μπορούσαμε να διαμορφώσουμε την περίοδο χρηματοδότησης Αυτό έχει να κάνει λίγο και με το κριτήριο επιλεξιμότητας που έθεσε πριν ως ερώτηση ο συνάδελφος. Και μια άλλη ερώτηση. Ο κύριος Κέλλη προηγουμένως ανέφερε τον περιορισμό των τριών ετών διάρκειας. Μετά τι γίνεται μετά τα τρία χρόνια. στα πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αυτής της ανταλλαγής εμπειρίας, αυτών των σχεδίων, αυτής της δημιουργίας δικτύων. Για την πρώτη ερώτηση του κυρίου Αλμπρίχτ ή του κυρίου Βανίστερόη, αν κατάλαβα καλά, τι σημαίνουν αυτά τα ποσά μοχλός. Μα είναι η πραγματική επίδραση, είναι αποδεδειγμένο δηλαδή, μπορεί να φέρει η γραμματεία μία απόδειξη, να σας αποδείξει δηλαδή πώς επηρεάζουν τα κονδύλια του Interact 3S επί συνολικά των κονδυλίων των διαπεριπεριακών προγραμμάτων. Πριν σας ανέφερα 7, 7 εκατομμύρια ευρώ του κάτρωσε του 4 σε, συγγνώμη, σε τέσσερα σχέδια πρόκειται για σχέδια κεφαλαιοποίηση. Ζητούμε να υπάρχουν διαχειριστικές αρχές των περιφερειακών προγραμμάτων γύρω από το τραπέζι και αυτό καθιστά τα προγράμματα πολύ πιο λειτουργικά όταν πρέπει να περάσουμε από την ιδέα στην απόφαση. Αυτά τα 7 εκατομμύρια ευρώ μας επέτρεψαν να επιδράσουμε 574 εκατομμύρια ευρώ μέσω των καλών πρακτικών για αυτά τα σχέδια ε, υπάρχει και ένα άλλο που πρέπει να το προσέξουμε είναι το B3 Regions που με 1,5 εκατομμύριο FEDER Interreg 4C ε, επηρέασε στην εφαρμογή στην εγκατάσταση μάλλον του Ιντερνετ στην Ήπεθρο. 470 εκατομμύρια ευρώ επέφεραν αυτές ε, επέφερε αυτή η εγκατάσταση. Υπήρξε λοιπόν αυτό το φαινόμενο μοχλός. Θα μπορούσε κανείς να υπολογίσει αυτό το φαινόμενο μοχλό. και να πει ναι εντάξει το ίντερνετ στην Ήπεθρο οδήγησε και στη δημιουργία καλών πρακτικών αλλά θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε αλλιώς το τελικό νούμερο. Εμείς ως, ως γραμματεία μπορούμε να σας φέρουμε πάντως τις αποδείξεις για τα πιο ορατά σχέδια. Ε, εντάξει, αλλά για τα μελλοντικά σχέδια δεν μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε αν δεν έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Τώρα για τις διάφορες περιόδους, η περίοδος 5 κολλάει περισσότερο με την περίοδο 3 από ότι με την περίοδο 4 και αυτό είναι λυπηρό. Τώρα αν οι προτάσεις της Κομισιόν τις οποίες προετοιμάζουν έρθουν στο τραπέζι και θα είχαμε και άλλους δύο στόχους, ένα στόχο ανάπτυξης και ένα στόχο συνεργασίας, θα είχαμε τότε μία αναβάθμιση της συνεργασίας και από 2,5% θα περνάγαμε στο 7% όπως το λέει η κυρία Σάντσε Σμιτ στην έκθεσή της. Διότι ξέρετε, ερωτήθη για το πώς μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση, μα για να καλύψουμε τη ζήτηση πρέπει να αυξήσουμε τον προπολογισμό. Θα μπορούσαμε να έχουμε λοιπόν μια συμπερίληψη, μια νέα συμπερίληψη Interreg Interact που ξέρετε ότι το Interact αποτελεί μοχλό όλων των διαπεριφερειακών προγραμμάτων. Δεν κατάλαβα όλες τις ερωτήσεις του κυρίου Κέλλη για την ε, στρατηγική 2020 και για τα ποσοστά σύγκλησης και ποσοστά ανταγωνισμού. Μπορείτε να μου επαναλάβετε την ερώτηση για να μην σας απαντήσω άσχετα πράγματα. Το ερώτημά μου ήταν αν τα προγράμματα σχεδιάστηκαν για να συνάδουν με τη στρατηγική του 2020, τότε τι λόγο έχουν να ολοκληρώνονται μετά από 36 μήνες. Το είπε και η κυρία Σάντσες, κάτι παρόμοιο είπε και αυτή. Αυτό ήταν το ερώτημά μου. Εφόσον τα προγράμματα αυτά συμβάλλουν στην εφαρμογή της ε, στρατηγική για το 2020, γιατί να ολοκληρώνονται μετά από 36 μήνε, όταν το 2020 δεν ολοκληρώνεται παρά μόνο με το πέρα του έτους του 2020. <coughs> Θα προσπαθήσω να απαντήσω. για μας Επιτροπή Παρακολούθησης και Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φανερό ότι όταν κάνουμε την την τον αναπρογραμματισμό του προγράμματος Μακνό θα έπρεπε να ε, συμπεριλαμβάνεται και το Smart, το Green και τα λοιπά, δηλαδή ό,τι θέτει η συνθήκη της Λισαβόνας. Είναι απόλυτα νορμάλ να τα συμπεριλάβουμε όλα αυτά ως διάσταση και στρατηγικούς στόχους. Έχουμε θεματικά δίκτυα και ανταλλαγές που αποφασίσαμε να περιορίσουμε στη διάρκεια. Γιατί? Διότι αυτό το οποίο φοβόμασταν ήταν να δημιουργήσουμε μία ομάδα που όπως μία επιτροπή αρχίζει και διαλύεται ε, μέσα στο χρόνο και ξεχνιέται. Θέλαμε εμείς ένα περιορισμένο διάστημα οι πόλεις οι οποίες συνεργάζονται να καταλήξουν σε αποτελέσματα και σε συγκεκριμένα τοπικά σχέδια δράσης. Αυτό είναι, το, αυτός είναι ο λόγος της διάρκειας. Η σύνδεση με το 2020 όπως και προηγουμένως η σύνδεση με τη Λισαβόνα. Η θεματική πρόκληση, τα μεγάλα θέματα, οι μεγάλες προτεραιότητες της στρατηγική 2020, δηλαδή εμείς προτείνουμε στους υποψήφιους να έχουν σχέδια τα οποία κολλάνε μεταξύ τους και με τη στρατηγική 2020. Αυτό είναι το νόημα. Θελήσαμε λοιπόν στα τέλη των 36 μηνών να έχουμε τελειώσει τελικά σχέδια, τοπικά σχέδια δράσης, συστάσεις οι οποίες είναι εφαρμόσιμες. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι σε 18 μήνες, γιατί σε ένα χρόνο είναι πολύ λίγο, σε 18 μήνες, να κάνουμε μία μελέτη online, να θυμίσουμε, να, καλέσουμε όλες αυτές τις πόλεις, οι οποίες σύναψαν ένα συμβόλαιο τοπικής συνεργασίας. Τι κάνατε, Είπατε πριν από 1,5 χρόνο ότι εγκρίνατε τα σχέδια, έχετε και τη χρηματοδότηση. Ποια είναι η πραγματικότητα, όλοι χρειαζόμαστε αυτού του είδους τη δουλειά. Εγώ συνεχίζω για τις απαντήσεις σε άλλες ερωτήσεις που ετέθησαν. Υπάρχουν κριτήρια για να απαντήσουμε στον κύριο Γουαρό σχετικά με τη χρηματοδότηση των σχεδίων. φυσικά η επιλεξιμότητα δημόσιος φορέας 4D4C ε, και για το Ουρμπακ το οποίο συνεργάζεται με τις πόλεις. Μετά πρέπει να είναι κανείς ο οργανισμός, ε, δημόσιος φορέας. Υπάρχουν μετά και άλλα κριτήρια. Έχουμε συνεργασίες οι οποίες ε, δεν πρέπει να είναι πολύ κοντινές στο Ιντερεκ 4C πρέπει να έχουμε εταίρους από τις τέσσερις γωνιές της Ευρώπης. Μετά έχουμε ποιοτικά κριτήρια διαχείρισης, επικοινωνίας, σχεδίου δράσης, ακρίβειας κλπ τα οποία τα έχει επεξεργαστεί η Γραμματεία και τα έχουν εντεχθεί τα κράτη-μέλη. Αν τα νησιά μπορούν να έχουν πρόσβαση φυσικά. Και τα νησιά βέβαια δεν έρχονται συχνά διότι η απόσταση μπορεί να είναι ένας παράγοντας που τις μειώνει ως προς την εγκύτητα στο κέντρο πληροφόρησης Άρα γίνονται δεκτά τα νησιά. Τα έχουμε και στο Interreg 4C. Τώρα για το πόσο έχουμε προχωρήσει, εμείς έχουμε δεσμεύσει τα όλα, σχεδόν όλα τα ποσά, τα δύο τρίτα έχουν ήδη αποφασιστεί και έχουμε μόνο 100 εκατομμύρια ευρώ για τα οποία ακόμη δεν έχουμε αποφασίσει. αλλά κατατέθηκαν 355 σχέδια, 4.000 εταίροι που έχουν καταθέσει δηλαδή, τα οποία τα εξετάζουμε. Πρέπει να αποφασιστούν από τα κράτη-μέλη στα τέλη πέτωση του χρόνου. Συνολικά δηλαδή, τα κονδύλια του Interreg 4C ε θα δεσμευθούν φέτος και για τα νέα σχέδια θα πρέπει να περιμένουμε πια το 2014. Όμως, για το ΡΥΠ έχουμε ένα 4B Καραϊβική, ελπίζω ότι αυτό είναι το σωστό όνομα, ε, έχουμε εκεί κονδύλια και μετά από 7 χρόνια δουλειάς θα πρέπει να συζητήσουμε για να δούμε προς ποια κατεύθυνση πηγαίνετε εσείς για το σχέδιο Interreg ε, Καραϊβική, για την κυρία Σάντσε Σμιθ, η οποία η ίδια έχει συμβάλει ιδιαίτερα στο να δώσει απαντήσεις στα διάφορα προβλήματα, ε, απαντώ ότι η επιτυχία έγκυται στο ποσοστό παρέμβασης. και για να μπορέσει κανείς να αρχίσει να συμπληρώνει τέτοιου είδου ερωτηματολόγια στα αγγλικά πρέπει κανεί να έχει πολλά κίνητρα. Ασχολούμαστε ε, με μειονεκτικές περιοχές, ξεπεσμένες ε, περιοχές, βιομηχανικές ξεπεσμένες περιοχές και όταν καλούμε κάποιον και του λέμε έλα να κάνει συνεργασία, ε, πρέπει να του δώσεις κάτι το οποίο να λειτουργεί ως αντιστάθμισμα, το οποίο να δικαιολογεί δηλαδή και όλες τις πρακτικές, τις γραφειοκρατίες κτλ. Μία από τις απαντήσεις επίσης της κυρίας Μία από τις απαντήσεις της κυρία Σάντσες Σμιτ ε, σχετικά με αυτό το αίσθημα πίεσης ε, Ε, ε, αφορά στον προϋπολογισμό ο οποίος καλύπτει μόνο μέρος της ζήτησης και πρέπει να επικοινωνούμε καλύτερα και να λέμε ότι ακόμη και όταν κανείς είναι επιλέξιμος ε, για ένα πρόγραμμα δεν θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις οι οποίες δεν είναι καλά ζυγισμένες πριν έρθει σε επαφή με, τα γραφεία επαφής. Δεν αρκούν βέβαια τα τέσσερα γραφεία, χρειάζεται και υποστήριξη των κρατών. Μερικές φορές τα κράτη αισθάνονται μηχανία στο να φιλτράρουν τους ε, ίδιους τους, τους υπηκόους. Τέλος πάντων, θα τα καταφέρουμε. Εμείς βελτιώνουμε το ποσοστό επιλεξιμότητας. Πέρασε από 80% στο 86% με την ε, επικοινωνία κάνουμε διάτερες, ε, έχουμε διάτερες πετυχίες και το 4 σε είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά στην ανταγωνιστικότητα και ξέρετε και το πρόγραμμα για την έρευνα δεν έχει μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχίας από ότι το δικό μας. και έχουμε αυξήσει τα ποσοστά. Αλλά ε, η αύξηση αυτή δεν είναι τόσο σημαντική. Μέχρι τώρα μπορεί η Επιτροπή να αποφασίσει κάτι διαφορετικό έχουμε μια διαφορετική διαδικασία επιλογής του διαγωνισμούς. Υπάρχει μια σοβαρή διαφορά. Κανένας δεν ε, βγάζει λεφτά ερχόντα, ερχόμενος να δουλέψει στην, ε, στο Ουρμπακτ. Δεν χρηματοδοτούμε, δεν χρηματοδοτούμε τα τοπικά σχέδια δράσης. Επομένως, η ελκυστικότητα, η χρηματική είναι μηδενική. Και αυτό είναι σημαντικό για τον αριθμό των υποψηφίων που έχουμε. Έχουμε όμως ε, μία συζήτηση ε, που συνεχώς ανακύπτει όταν μας λένε ότι για παράδειγμα μπορούμε με αυτό το διαγωνισμό να δημιουργήσουμε 15 δίκτυα, αλλά εμείς τελικά μπορεί να έχουμε μόνο 13 δίκτυα πραγματικά καλής ποιότητας ε, και να... Επομένως, δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι η απάντηση είναι ας αυξήσουμε τον προπολογισμό και ας χρηματοδοτήσουμε όλους τους υποψηφίους. Αν θέλουμε να αυξηθεί η ποιότητα, να ανεβεί ο πύχης, πρέπει να κάνουμε μία επιλογή και νομίζω ότι αυτό είναι δυνατό. Βέβαια, τότε βρισκόμαστε σε επίπεδο περισσότερο πιλωτικών προγραμμάτων ε, που δείχνουν ότι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα τα οποία όντως ε, ε, αποτελούν πρόοδο. Αυτή είναι η άποψη της Επιτροπής Παρακολούθησης, ότι αυτή, το, αυτό το ζήτημα της αριστείας ήταν κεντρικό ζήτημα στην επιλογή των προγραμμάτων κατά τη διάρκεια των διαγωνισμών. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό το ε, βασικό ε, ζήτημα της σχέσης ε, με τις διαχειριστικές αρχές που ανέφερε ο κύριος Όλμπριχτ. Ναι, ήταν πολύ σημαντικό για το Ουρμπακτ. Δεν έχουμε κανέναν αυτόματο διαρθρωτικό σύνδεσμο με τις διαχειριστικές αρχές. Ένα τοπικό σχέδιο δράσης ε, καταρτίζεται σε ένα τοπικό επίπεδο μπορεί να χρηματοδοτηθεί ή όχι από το επιχειρησιακό πρόγραμμα αναλόγως με το αν έχουν ένα κεφάλαιο στον προπολογισμό τους για τα ζητήματα urban ε, ή αν υπάρχουν ακόμη κονδύλια διαθέσιμα ή αν υπάρχει κάποια ε, συνάφεια, εν πάση περιπτώσει, πολιτική με την πόλη που παρουσιάζει ένα πρόγραμμα. Τώρα, η σχέση με τις διαχειριστικές αρχές είναι πραγματικά βασικό ζήτημα για μας για τη συνέχιση τέτοιου είδους προγραμμάτων. Θα ήθελα κάτι ακόμη να προσθέσω ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε τη χρηματοδότηση, τη δυνατότητα χρηματοδότησης και τη γνώση των αστικών πολιτικών. Πολλές διαχειριστικές αρχές χρηματοδοτούν προγράμματα που παρουσιάζουν οι πόλεις, αλλά δεν έχουν κανένα όραμα για, το, για, ε, για, τις, πόλεις τους, που είναι για μένα ένα αρκετά σημαντικό ζήτημα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, που είναι το πρόβλημα ε, της ε, ενίσχυσης των τεχνικών υποδομών, να υπάρχει μια πραγματική αστική στρατηγική. Γι' αυτό μιλάω για το Urbact. Για μένα είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά την επόμενη περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τροβινή. Τώρα να δώσουμε το λόγο στους δύο εμπρογνώμονες της Κομισιόν. Ο κύριος Κόρς uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Κομισιόν συμμερίζεται τις αναλύσεις και τις ε, απόψεις που παρουσίασε ο κύριος Δρουμπινή το Urbact όντως αποτέλεσε ένα πρόγραμμα διασύνδεσης πόλεων πολύ επιτυχές που δημιουργήθηκε ως ε, εργαλείο για να ανταλλαγούν εμπειρίες μεταξύ πόλεων που συμμετέχουν στην ε, κοινή πρωτοβουλία της Urbact, στην ε, εκπόνηση του δικτύου των πόλεων του Urbact και ο αριθμός των πόλεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό μετά την ε, τρίτη ε, πρόσκληση ε, διαφέροντος θα είναι περίπου 440 πόλεις. Υπήρξε ένα θέμα για το γιατί δεν υπάρχει επαρκή σύνδεση μεταξύ των, του προγράμματος δικτύωσης και των βασικών mainstream επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ότι τα κονδύλια για τα βασικά προγράμματα αποφασίζονται από πολύ καιρό πριν. Και οι καλές ιδέες που εκπονούνται τώρα μπορεί να μην μπορούν να χρηματοδοτηθούν γιατί δεν υπάρχουν κονδύλια πια διαθέσιμα. Παρ' όλα αυτά, με το Urbact μπορούμε να είμαστε περήφανοι γιατί πραγματικά έχουμε φτάσει σε μια πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων δικτύων πόλεων και των διαχειριστικών αρχών. Και αυτό έγινε σε θελούσια βάση, σε θελούσια, ε, με θελούσια συμμετοχή των διαχειριστικών αρχών. Και πολλέ ιδέε που εκπονήθηκαν στα πλαίσια του Ούρμπακτ ήταν πολύ επιτυχημένε. Η Κομισιόν επέλεξε έναν αριθμό δικτύων στα πλαίσια του Fast Track και του σχετικού δικτύου. Αυτά τα δίκτυα Fast Track ε, έλαβαν κάποια υποστήριξη από την Κομισιόν Κάποια έλαβαν και υποστήριξη από το Κοινοβούλιο. Ένα από τα δίκτυα αυτά είναι το UNIC, το οποίο αποτελείται από πόλεις που εξαρτώνται από τον τομέα της κεραμικής και το Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει ενεργά. Έχει στηρίξει τη δουλειά αυτού του δικτύου. Και επίσης ένα άλλο ε, επιτυχημένο δίκτυο Fast Track, το Milo για την ε, ε, ενσωμάτωση των μεταναστών. Μόλις ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αυτό, είδαμε ότι στα πλαίσια του δικτύου υπήρχαν πάρα πολλές καλές ιδέες, τις οποίες υιοθέτησε η Διαχειριστική Αρχή. Και αυτό είναι, συμβαίνει και, για την Πορτογαλία, και στην Πορτογαλία, γιατί ένα τμήμα του δικτύου Mile είχε να κάνει με την προώθηση της ένταξης των μεταναστών μέσω κάποιων ε, ορχιστρών, μέλη των οποίων ήταν ε, τα παιδιά των ε, μεταναστών, των οικογενειών των μεταναστών. Και αυτό έχει συμβεί και σε άλλες πόλεις, το έχουμε αντιγράψει. Ο κύριος Ντουρμπινή επίσης μίλησε για το για τις νέες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, για τις νέες προτεραιότητες επίσης για το 2020 ε, θα πρέπει να απαντήσουμε και εμείς και επίσης θέλουμε να ξεκινήσει το πιλωτικό εγχείρημα ε, μιας ανταλλαγής ε, ε, εκλεγμένων τοπικών συμβούλων ή μελών της τοπικής αυτοδιοίκησης ως follow-up, ως συνέχεια του πολιτικού προγραμμά, προ, πιλωτικού προγράμματος Εράσμους για τους ε, ερετούς άρχοντες που στηρίζει και το Κοινοβούλιο. Βεβαίω θα χρησιμοποιήσουμε, θα κεφαλοποιήσουμε την εμπειρία του Ούρμπακτ όταν θα υποβάλουμε τη νέα πρόταση για το νέο προγραμματική περίοδο για την πολιτική συνοχή και βεβαίω θα προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που έχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να συνεχιστεί η επιτυχή συνεργασία του δικτύου των Ευρωπαϊκών Πόλεων. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ο κύριος Βενινό έχει τώρα το λόγο. Merci, Monsieur le Président. Euh, Ο Μισελ Λαμπλά ανέφερε όλες τις ευκαιρίες ε, της ε, διασυνοριακής συνεργασίας με το Interreg 4C, ε, όπως επίσης και τις προκλήσεις που θα πρέπει να δράξουμε σήμερα. Πρέπει όμως να σταθούμε σε κάτι εμφανές. Είναι το μόνο πρόγραμμα σήμερα στην Ευρώπη που επιτρέπει σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη να ανταλλάξουν τις πρακτικές τους, τα σχέδιά τους για να τα εφαρμόσουν στη συνέχεια σε πιο τοπικό επίπεδο και να μπορέσουν έτσι να, είναι, ευεργετηθούν ε, από τα κεκτημένα και τις εμπειρίες ορισμένων από αυτές τις περιοχές. Το σημείο που ανέφερε ο Μισελ Λαμπλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό ε, και είναι αυτό το οποίο λέει ότι νέες χώρες που μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον αυτοί που παρουσιάζουν τα περισσότερα σχέδια και ευεργετούνται από αυτήν την μεταφορά και ανταλλαγή εμπειρίας. Πρόκειται για ένα συνεκτικό στοιχείο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι λοιπόν μια πρώτη, ένα πρώτο επιχείρημα το οποίο σας αναφέρω υπέρ της επέκτασης και της συνέχισης αυτού του προγράμματος για το 2014-2020. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού συνδέεται με αυτό. Αν θέλουμε εμείς να συνεχίσουμε να εκμεταλλευόμεθα ε, ορισμένες ε, εμπειρίες πιο λειτουργικά, θα ήταν λογικό ο προϋπολογισμός της επόμενης περίοδου και αυτός να αυξηθεί. Σήμερα έχουμε δύο προτεραιότητες, Λισαβόνα και Γκέτεμποργκ, τις ανέφερε ο Μισελ Λαμπλά. Στα πλαίσια του Youth 2020, Ευρώπη 2020, θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Αν μπορούμε δηλαδή να έχουμε μία επέκταση του πεδίου προτεραιοτήτων και να δει το θέμα της διαχείρισης αλλά και το θέμα της διοικητικής και θεσμικής ικανότητας. Εδώ πρέπει να έχουμε ένα στοιχείο ανάκτησης ορισμένων και εκτιμένων μερικών περιφερειών οι οποίες σήμερα είναι ακόμη σχετικά ελληματικές θεσμικά και διοικητικά. Και αν θέλουμε εμείς ε, στην επόμενη γενιά διαπεριφερειακής συνεργασίας να καταπολεμήσουμε αυτό το φαινόμενο, θα πρέπει να επιταχύνουμε στα θεματικά ζητήματα τα οποία υποστηρίζονται στο τωρινό πλαίσιο του Interreg 4C. Θα έχουμε στοιχεία τα οποία πιστεύουμε ότι είναι σημαντικά και πρέπει να τα αναπτύξουμε και όσον αφορά στο θέμα της επικοινωνίας εμείς έχουμε ως στόχο του χρόνου την άνοιξη να έχουμε μια μεγάλη διάσκεψη που θα επιτρέψει στους πρωταγωνιστές της διαπεριφερειακής συνεργασίας να έρθουν σε επαφή με τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες για να τονίσουν ορισμένα αποτελέσματα τα οποία μπορούμε κάλλιστα ε, σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς, στρατηγικής ε, και καινοτομίας. Έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να τονιστούν και να αποδείξουν και την προστιθέμενη αξία του προγράμματος. Επίσης, μετά από την απόφαση που λήφθη στο Όσλο σε μια επιτροπή παρακολούθησης, προσπαθήσαμε να τονίσουμε σε επίπεδο προγράμματος συνολικά όλα τα απορίσματα τα οποία μπορούμε εμείς ε, να έχουμε ε, αναλύοντας την εμπειρία ορισμένων από αυτά τα network. Όταν θα έχουμε μία κριτική μάζα σχεδίων μέσω που θα μας έρθουν μετά από πολλά δίκτυα, τότε οι εμπειρογνώμονες θα μπορέσουν να μας καταδείξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα που μπορούν να παράγουν αυτές οι περιφέρειες ως εξέλιξη των πολιτικών τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και τον δεσμό που ανέφερε ο κύριος Όλμπριχτ δεσμό μεταξύ προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης και συνεργασίας και προγραμμάτων συνεργασίας. Είναι θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν συνολικά τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες. Είτε είναι περιβαλλοντικά, είτε οικονομικά, είτε έχουν σχέση με την αλλαγή του κλίματος. Χρειάζονται ανάπτυξη ενός νέου ε, μέσου συνεργασίας το οποίο δεν θα πρέπει να αποτελεί απλώς προσθήκη να λειτουργεί προσθετικά στις προσπάθειες που γίνονται σήμερα αλλά θα έπρεπε να αποτελούν στοιχείο, νέο στοιχείο μέσα στις στρατηγικές. Μπορεί να είναι αυτός ευσεβής πόθος. αλλά έχουμε την πεποίθηση ότι η συνεργασία αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της περιφερειακής ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν εμείς να βρούμε έναν καλύτερο τρόπο για να διασφαλίσουμε αυτή τη σχέση. Και ό,τι έχουμε ως και στα προγράμματα συνοχής και συνεργασίας να περάσει και στα αναπτυξιακά προγράμματα των περιφερειών. Τελευταίο, έχουμε τρία προγράμματα συνεργασίας ε, διεθνική συνεργασία σήμερα μέσα στα πλαίσια του κεφαλαίου 4B, Καραϊβική, Ινδικός ωκεανός, Αζόρες, Μαδέρα και Κανάρια νησιά. Να λαμβάνοντα υπόψη δηλαδή και τη γεωγραφική εγκύτητα. Σμιτ η κυρία Σάντσε Σμιτ μπορεί τώρα να κλείσει τη συζήτηση. Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους κυρίους Λομπλέν και Τζουμπινί Νομίζω ότι και στις δικές τους παρεμβάσεις αλλά και στις ερωτήσεις των συνοδέλφων και στα λόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είδαμε το, τη σημασία ε, αυτής της διασυνοριακής συνεργασίας. Είμαστε πεπισμένοι νομίζω ε, για την υποστήριξη που μπορεί να ε, προσφέρει η διασυνοριακή συνεργασία, πώς μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της ε, εδαφικής συνεργασίας και συμφωνώ απολύτως με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής που ανέφερε την αναγκαιότητα ύπαρξης ε, γεφυρών μεταξύ όσων ήδη ε, υφίστανται και των προγραμμάτων που θα προβλεφθούν. Νομίζω ότι πολύ συχνά πολλοί εξημών αναφέρουν ότι η ευρωπαϊκή πολιτική και συγκεκριμένα η περιφερειακή πολιτική εμπροκειμένου πρέπει να ε, καταδείξει την προστιθέμενη αξία της. Μιλάμε λοιπόν για κάτι πολύ συγκεκριμένο, ε, πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Βεβαίως οι μεγάλοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 πρέπει να ληφθούν υπόψη σε όλες τις πολιτικές μας, αλλά μπορούμε και επιτόπου να δείξουμε πόση προστιθέμενη αξία μπορούμε να επιφέρουμε ε, στην καθημερινή ζωή των πολιτών και στην οικονομική ζωή Επίσης ε, αναφερθήκατε πολύ για τα, στα θέματα της επικοινωνίας και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να να υπάρχει επικοινωνία μέσω των ε, περιφερειακών προγραμμάτων και είναι πολύ σημαντική και η γνώση. Τίποτε δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εμπειρία. Έχουμε λοιπόν ένα καθήκον να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις γνώσεις και όλες αυτές τις ε, εμπειρίες μέσω της ανταλλαγής ε, καλών πρακτικών, γιατί η περιφερειακή πολιτική είναι μια πολιτική επενδύσεων και έχει, ένα στόχο, έχει ως στόχο την ε, κοινωνική, οικονομική και τοπική ανάπτυξη. Το να δείξουμε λοιπόν πώς θα φτάσουμε σε αυτήν την ανάπτυξη ε, είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό. Και στην έκθεση την οποία έχω την τιμή να ε, συντάξω ζητήθηκε μια ενίσχυση της συγκεκριμένης συνεργασίας και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι υπόλοιποι κανονισμοί και οι μελλοντικοί κανονισμοί, ε, ακόμη και αν δεν τα καταφέρνουμε να, επιτύχουμε το 100% ε, όλων όσων ε, ε, είχαμε ζητήσει. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε την, ε, τον τριπλασιασμό ε, ορισμένων κονδυλίων και νομίζω ότι αυτό αποτελεί μια ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας πολύ σημαντική και δείχνει τη σημασία του, του, της συνεργασίας των διαφόρων εταίρων στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας. Όσον αφορά το θέμα των τοπικών εκλεγμένων, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεργασία τους για την τοπική διακυβέρνηση και Επίσης, μας φέρνει πολύ πιο κοντά στους στόχους μας και στην πραγματικότητα αυτής της περιφερειακής πολιτικής. Νομίζω ότι είναι παιδαγωγικής φύσεως σχεδόν το θέμα. Θέλουμε πραγματικά να δείξουμε τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτύχει. πολύ. Ε, Επιτρέψτε μου πριν ολοκληρώσετε κύριε Πρόεδρε να θυμίσω ότι μετά τη λήξη της συνεδρίασης θα έχουμε ένα μικρό κοκτέιλ έξω από την αίθουσα. Η οικειότητα βοηθάει στην ανταλλαγή των καλών πρακτικών γενικότερα. Καλά τον κύριο Ντραμπίνι. Ε, να σας θυμίσω ότι μια επιτροπή, ένα, ένα κλιμάκιο της επιτροπής μας θα επισκεφτεί την ε, Βόρεια Ελλάδα ε, από αύριο κιόλας και θα έχουμε κάποια συμπαράσματα τα οποία και θα σας φέρουμε μετά τις διακοπές. Καλά να περάσετε. Η επόμενη συνάντηση είναι στις 19 ε, Σεπτεμβρίου ε, το φθινόπωρο.